Nous reprenons Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Να σας ενημερώσω ότι συνεδρίασαν οι συντονιστές αμέσως μετά την πρωινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής ε, και έλαβαν ε, μια σειρά αποφάσεων. Θα λάβετε τα πρακτικά στο ηλεκτρονικό στοιχειοδρομείο των αποφάσεων των συντονιστών και επίσης ε, για τις διάφορες εκθέσεις που θα ε, μπουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αποφασίσαμε να κρατήσουμε τους ίδιους ε, εισηγητές και συνεισηγητές ε, εφόσον υπάρχει επανεκλογή και για όσους δεν έχουν επανεκλογή θα τηρήσουμε τις πολιτικές ισορροπίες που είχαν βρεθεί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία για να ανανεώσουμε τους εισηγητές και συντάκτες γνωμοδότησης. Επίσης, αποφασίσαμε να καλέσουμε τον Επίτροπο Μπαρνιέ για να διαμορφώσουμε μια πιο συγκεκριμένη άποψη των συνεπειών μιας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, ενός no deal που σίγουρα θα γίνει. Σίγουρα και η δική μας Επιτροπή θα επηρεαστεί τα μάλα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποκομίσουμε μια πιο σαφή εντύπωση για το τι θα συμβεί μετά την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, μετά από ένα no deal που είναι σχεδόν σίγουρο. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο ηλεκτρονικό στοιχειοδρομείο ως προς τις αποφάσεις των συντονιστών. Συνεχίζουμε λοιπόν με την παρουσίαση μιας μελέτης που θα μας παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα ο τμήματάρχης της μονάδας έρευνας τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του και να σας υπενθυμίσω ότι εκτός από τους ε, ε, εμπειρογνώμονες που έχουμε στη Γραμματεία και στις πολιτικές ομάδες, έχουμε μία μονάδα έρευνας που συνδράμε την Επιτροπή μας. Και μάλιστα αυτή η μονάδα είναι αρμόδια για την ε, εκπόνηση ή ανάθεση εκθέσεων για θέματα που μας ενδιαφέρουν με βάση ένα εξάμηνιαίο πρόγραμμα εργασιών που έχουμε προεγκρίνει. Δύο διοικητικοί υπάλληλοι παρακολουθούν μάλιστα το έργο της Επιτροπής Ρέγγι. Ο τμετάρχης ο κύριος Ιωάννης Λίτζελμαν, που είναι παρόν. Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης που είχε ζητήσει η απερχόμενη Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το θέμα είναι ευρύτατο βέβαια, αλλά έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα και πιστεύω ή ελπίζω τουλάχιστον θα μας επιτρέψει να ενημερωθούμε καλύτερα και κυρίως τα νέα μέλη για τα θέματα της πολιτικής συνοχής και της προτεραιότητές της. Έτσι θα είμαστε πιο κατατοπισμένοι και θα συνειδητοποιήσουμε τη θέση που έχει η συνοχή στις γενικότερες συζητήσεις ε, που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη μελέτη θα μας παρουσιάσει ο κύριος Κάλλος Μέντες από το Πανεπιστήμιο Στράχκλιντ του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δώσω όμως πρώτα το λόγο στον κύριο Μέντες για ένα τέταρτο. Μάλλον στον κύριο Λίτσελμαν για ένα, για ένα τέταρτο πρώτα, μετά στον κύριο Μέντες για άλλο τέταρτο και θα ακολουθήσει η συζήτηση στην οποία πιστεύω θα υποβάλλουν τις απορίες τους στα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων που μου δίνετε την ευκαιρία πριν την παρουσία της μελέτης να σας παρουσιάσω εν συντομία το τμήμα πολιτικής ε, που δημιουργήθηκε μαζί με άλλα το 2004 για να συνδράμει το έργο των γραμματιών των επιτροπών στα θέματα έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη. Όλε οι επιτροπέ έχουν ένα τμήμα πολιτική που συνεργάζεται μαζί του, όπω βλέπετε στη διαφάνεια. Και η... ο καθρέφτη αυτού του τμήματο πολιτική ε, είναι η διοικητική διάρθρωση τη γραμματεία. Σε ό,τι αφορά τη δική σα επιτροπή, ε, εμείς καλύπτουμε ταυτόχρονα την Επιτροπή Άγκρη, Αλίας, ε, Βιομηχανίας και Πολιτισμού. Όπως σας είπα, παρέχουμε υπηρεσίες έρευνας ε, και εμπειρογνωμοσύνη σε κοινοβουλευτικά σώματα, όχι σε μεμονωμένους ευρωβουλευτές. Και αυτή είναι, η διαφορά μεταξύ του τμήματος πολιτικής και της μονάδας μελετών IPRS, που εκπονεί εκθέσει μετά από συγκεκριμένα αιτήματα μονομένων ευρωβουλευτών. Αυτή είναι η ειδοποιό μα διαφορά από την υπηρεσία EPRS. Εμεί προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στι προτεραιότητε τη Επιτροπή και στη διαδικασία λήψη αποφάσεών τη. Για παράδειγμα, θέλουμε να διαλευκάνουμε τεχνικέ ε, και νομικέ ε, ε, θέσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου και το κάνουμε αυτό με τη διαχείριση του προπολογισμού και με συνεχείς και άμεσες επαφές με τους ερευνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρουμε χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση προσανατολισμένη προς τη δράση. Στόχο έχει να σας δώσουμε κάποια σενάρια ή επιλογές πολιτικής ή κάποιες συστάσεις πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο καθημερινό σας κοινοβουλευτικό έργο. Επίσης, παρέχουμε πραγματογνωμοσύνη που ε, περιλαμβάνεται στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ε, στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής ΡΕΓΚΙ. Επίσης, ε, επειδή στις έρευνες μας μερικές φορές αγγίπτουμε και σε ευαίσθητα πολιτικά θέματα, επιμένουμε στην διαφάνεια, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία. Και αυτό το κάνουμε με οργάνωση διαγωνισμών που είναι δημόσιοι, διαφανείς και επίσης έχουμε πολύ σαφή και αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές ό,τι αφορά την επιλογή των συμβαλωμένων μερών. Και αυτό γίνεται από μια επιτροπή με μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης χρησιμοποιούμε διαδικασίες αξιολόγηση ομοτήμων και έχουμε και ειδικά εργαλεία για να αποφεύγουμε τις αντιγραφές Μάλιστα, την πραγματογνωμοσύνη μας τη δίνουμε με, διάφορες, ε, με διάφορους τρόπους. Καταρχήν έχουμε σύντομες μονοσέλιδες, δισέλιδες ε, σε ενημερώσεις, ε, πιο εκτενείς ενημερώσεις ή πιο ευρυθείς ενημερώσεις, 11-36 σελίδες, που είναι το βασικό τμήμα των της, προσφορ... της συνεισφοράς μας. Όλες οι μελέτες μας εκπονούνται στα αγγλικά και επίσης δημοσιεύονται μόνο στα αγγλικά. Και αυτό οφείλεται στις περιορισμένες δυνατότητες μετάφρασης που έχουμε. Γιατί δίνεται προτεραιότητα στη μετάφραση των νομοθετικών κειμένων. Δεν προλαβαίνουμε να μεταφράσουμε και τις έρευνες. Τώρα, αν κάποια συγκεκριμένη μελέτη σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, μπορούμε να τη μεταφράσουμε σε μερικές άλλες γλώσσες, αλλά όχι συστηματικά σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ε, αλλά πολύ συστηματικά δίνουμε, προσφέρουμε ε, συνόψεις ε, για τις εκθέσεις μας και σε άλλες γλώσσες. Επίσης οργανώνουμε και εργαστήρια και πάνελ ε, εμπειρογνωμόνων και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά σας τα ε, δίνουμε με σύντομες ενημερώσεις. Μάλιστα, εμπειρογνωμοσύνη ε, την αντλούμε είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσωτερικά και έχουμε μόνο δύο διοικητικούς υπαλλήλου που παρακολουθούν το κάθε τομέα εμπειρογνωμοσύνης, οπότε έχουμε περιορισμένα μέσα, κάτι που σημαίνει ότι οι περισσότερες μελέτες ανατίθενται εξωτερικά μέσα από διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών. Αυτές οι διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών είναι πολύ άρτιες γιατί μας επιτρέπουν να έχουμε επαφή με ειδικού εμπειρογνώμονες, ειδήμονες για κάποια θέματα, αλλά το αρνητικό τους σημείο είναι ότι είναι χρονοβόρες διαδικασίε και ξεκινά από μια απόφαση των συντονιστών να εκπονηθεί μια μελέτη. Μετά γίνεται ο δημόσιος διαγωνισμός που η διαδικασία αυτή κρατάει 1,5 με 4 μήνες. Μετά θα πρέπει να δώσουμε ε, το χρόνο στους ερευνητές να εκπονήσουν τις μελέτες τους, 2 με 6 μήνες και μετά έχουμε τον ποιοτικό έλεγχο και ε, αν χρειαστεί και τη μετάφραση κάτι που κρατάει ένα με δύο μήνες. Οπότε η όλη διαδικασία κρατάει από 4 μέχρι 12 μήνες από την απόφαση των συντονιστών μέχρι να φτάσουμε στην παρουσίαση της συγκεκριμένης έκθεσης στην Επιτροπή. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι όλες μας οι μελέτες είναι δημοσίως προσιτές, είναι δημόσια πρόσβαση εξασφαλισμένη και μάλιστα έχουμε ε, τις εκθέσεις μας και στην, στη σελίδα της Ρέγγι, στο ίντρανετ ε, και ε, είμαστε, βρισκόμαστε και στο Twitter και εκεί ε, εκδίδουμε ενημερωτικά δελτία, αλλά έχουμε και ε, ε στη βιβλιοθήκη τις εκθέσεις μας και τις μελέτες μας σε έγγραφα. Τώρα, εν συντομία να σας πω τι κάναμε στο παρελθόν και ποιος είναι ο στόχος μας για το μέλλον. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία δώσαμε στην Επιτροπή Ρέγκη 36 εξωτερικές μελέτες για πολλά και διάφορα θέματα. Εδαφική διακυβέρνηση και πολιτική συνοχή, πολιτική συνοχή και στόχοι τη Συμφωνία των Παρισίων, πολιτική συνοχή και κρατικέ ενισχύσει και ούτω καθεξή. Επίση, οργανώσαμε εννέα εργαστήρια, workshops για το μέλλον της πολιτικής συνοχή, Πολιτική συνοχή και κλιματικέ αλλαγέ και εκπονήσαμε και μια σειρά άλλων μελετών και ενημερώσεων που μπορείτε να τις βρείτε στο ίντρανετ. Τέλος, ολοκληρώσαμε και τέσσερις μελέτες που θα δημοσιευτούν το 2019. Τη μία θα σας την παρουσιάσει αμέσως μετά τη δική μου παρουσίαση ο κ. Μέντες. Το θεματολόγιο της πολιτικής συνοχής για το 2019 μέχρι το 2024 πρόκειται για μια οριζόντια, όπως λέμε, μελέτη ε, και έχουμε και πιο συγκεκριμένα θέματα, τη διάσταση του φύλου στη, στην πολιτική συνοχή, το αστικό θεματολόγιο και την προβολή και επικοινωνία. Ένα θέμα που θα σας αναπτύξει ο κύριος Μέντες στα πλαίσια της μελέτης που εκπονήσαμε. Σε ό,τι αφορά το μέλλον. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μελέτης για το τι ε, θα προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κατάλογο μελετών για το 2020. Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνει αυτό. Και βασικός μας στόχος είναι ότι προβλέψουμε να είναι πλούσιο σε αποτελέσματα για εσά και να μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τι συνεισφορέ σα από όλε τι πολιτικέ ομάδε για το τι μελέτε να θέσουμε ω προτεραιότητα για τι αρχέ του 2020. Και με αυτά ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα. Merci Ευχαριστούμε πολύ. Και με την ευκαιρία να τονίσω και εγώ πώς εκτιμούμε τη δουλειά της ε, υπηρεσίας σας. Μελέτες εξαιρετικά χρήσιμες που ενισχύουν τη δουλειά της Επιτροπής μας και θα ζητήσω από τους συναδέλφους να διαβάσουν τη μελέτη αυτή γιατί ε, ο, αυτοί όπως και προηγούμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί μπορούν να μας βοηθήσουν να καταρτήσουμε καλύτερες προτάσεις ε, που έχουμε να σας κάνουμε ως τα τέλη Οκτωβρίου για να ανοίξουμε και νέους δρόμους, να βρούμε νέες ιδέες για το τι μπορεί να μας απασχολήσει στο μέλλον. Και τώρα λόγω στον κύριο Μέντες. το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε και κύριοι βουλευτές. Θέλω να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη ε, που έχουμε ε, διευθύνει από κοινού με τους συναδέλφους Μπάκλερ και Μάκ Μάστερ από το Πανεπιστήμιο του, του ΤΕΛ στην, ε, στις κατοχώρες. Πολύ σύντομα οι στόχοι και μετά τα, ε, οι έξι ομάδες στόχων και συστάσεων προκύπτουν από τη μελέτη. Επτά τομείς ε, που αφορούν ε, την πολιτική, την περιφερειακή και βάσει των ε, κανόνων του Κοινοβουλίου μας απασχόλησαν. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα όλες τις λεπτομέρειες, θα συνοψίσω και θα επικεντρωθώ περισσότερο στις συστάσεις, ιδίως αυτές που αφορούν το Κοινοβούλιο και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ένα από τα βασικά θέματα, από τα πρώτα βασικά θέματα, ήταν ε, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η απουσία ενός συγκεκριμένου πλαισίου για το στρατηγικό σχεδιασμό. Βεβαίως, τώρα έχουμε και το πρόγραμμα Ευρώπη 2020, που έχει και το CSF που έχουν συγκεκριμένους στόχους για αυτή την περίοδο, όμως πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή με τη συγχρηματοδότησή τη, που να μην είναι τυφλίω προ του ε, επιμέρου τελικού στόχου. Θέλουμε βεβαίω περισσότερη συνοχή σε όλα τα επίπεδα, αλλά και να υπάρχει ένα κοινό σκοπό για όλου του εμπλεκομένους σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή το στρατηγικό πλαίσιο επιτρέπει να οριστούν και να υλοποιηθούν στόχοι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως τα χαμηλότερα, με πιστή επιδίωξη των στόχων αυτών, σταθερή επιδίωξη των στόχων, Και βεβαίω η νέα ατζέντα για το 1924 δεν καλύπτει το θέμα αυτό. Το έγγραφο, όπω είπα, είναι πάρα πολύ ευρύ, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη έκφραση σε συγκεκριμένου τομεί. Η βασική σύσταση είναι το Κοινοβούλιο να καλλιεργήσει μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση που να επικεντρωθεί και στου τόπου και στου χώρου, ώστε η συνοχή να λαμβάνεται υπόψη τόπου, αλλά να υπάρχει ένα ουσιοδό, ε, ουσιαστικά μάλλον στρατηγικό επίπεδο όχι μόνο οι εδαφικές μελέτες αντικτύπου, που και αυτές είναι σημαντικές. Τώρα για την συνοχή των κονδυλίων. Απειλείται από τις νέες προτάσεις. Πολλοί είναι οι εταίροι που προβάλλουν το επιχείρημα ότι είναι κρίσιμη η σχέση της συνοχής με το CSF sin και την περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό σε επιχείρημα, αλλά πρέπει να δούμε και την αποχώρηση του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπέθρου από το κοινό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρξει μεταφορά λοιπόν από την πολιτική συνοχής προς κοινώς ε, διαχειριζόμενα προγράμματα. πρέπει να μην αλλάξει και αποδυναμωθεί η πολιτική προσέγγιση ως προς τον τόπο, τον χώρο. Θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες διαδικασίες και όχι κατακαιρματισμός της ε, προσέγγισης των ε, διαφόρων θεμάτων. Η Επιτροπή Ρέτζι στις εκθέσεις της περιλαμβάνει συχνά συστάσεις για το πώς θα πρέπει το Ταμείο Ανάπτυξης της Πέθρου να συνδυαστεί με τις διάφορες συστάσεις και την ενίσχυση των στόχων και να υπάρχει περισσότερος συντονισμός των κονδυλίων βάσει του πολιτικού στόχου 5. Πρέπει λοιπόν να επιδιωχθούν αυτές οι προτεραιότητες κατά τη διάρκεια των ε, τριμερών διαλόγων, αλλά και για να εξετάσουμε προσεκτικά την επίτευξη στόχων ε, στην ερχόμενη θητεία ιδίω. Για τις εταιρικέ σχέσεις. Βασικά υπάρχει το θέμα μετα... της σύγκρισης μεταξύ ε, συμμετοχικής και αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης η οποία με βάση τις διαβουλεύσεις γρήγορα και αποτελεσματικά να οδηγεί σε καρπούς, χωρίς να είναι αναγκαστικά και νομικού χαρακτήρα. Το Συμβούλιο έχει επιλέξει μια πιο γενικόλογη διατύπωση, μιλώντας για αρμόδιους εταίρους, για κώδικες συμπεριφοράς, ενώ το Κοινοβούλιο θέλει μια πιο καλά πλαισιωμένη και προσεκτικά καθορισμένη εταιρική σχέση. Υπάρχει περιθώριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τον κώδικα συμπεριφορά, να τον αναθεωρεί ετησίω, ώστε να υλοποιείται και στι εταιρικέ σχέσει προσεκτικότερα. Θα πρέπει να δούμε και τι ριζοσπαστικότερες προτάσει για την επέκταση των εταιρικών σχέσεων προ μια νέα κατεύθυνση, αλλά σε μια μελλοντική φάση. Το τέταρτο θέμα είναι η οικονομική διακυβέρνηση. Ε, η διεύθυνση των οικονομικών υποθέσεων. Εδώ παίζουν ρόλο το, οικονομικό, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, συγγνώμη, η αναχώραση τάση, η πολιτική συνοχή και την τελευταία περίοδο προγραμματισμού ενισχύθηκαν. Θέλουμε περαιτέρω ενίσχυση και στο μέλλον και η αρεσιμότητα καθώς και οι εξελισσόμενε, ε, οι ενεξελίξει μάλλον εντάσει μεταξύ του μέλλοντο των ιδιωτικών ταμείων και τη πολιτική συνοχή. Βασική μα σύσταση είναι να ακολουθήσουμε μια οικονομική διακυβέρνηση περισσότερο εδαφικού χαρακτήρα, δηλαδή να δούμε τι προτεραιότητε επενδύσεων των ε, χωρών με βάση τι αναχώρα εκθέσει, όπω εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο παράρτημα D, να δούμε ως το 2024 αυτή η εδαφική προσέγγιση πώς μπορεί να ε, υλοποιηθεί. Είναι βέβαια σύντομα σε έκταση τα έγγραφα που έχουν ετοιμαστεί, όμως μπορεί πιο εύκολα κανείς να κάνει τις συγκρίσεις μεταξύ των ε, προγραμμάτων αναχώρα και ούτως ή άλλως απότερος και γενικότερος ο στόχος της ε, διορθωτικής μεταρρύθμισης που χρειάζεται, της δομικής μεταρρύθμισης που χρειάζεται για συνοχή στι ε, περιφέρειες. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομικέ πολιτικέ πρέπει να λάβουν υπόψη την συνοχή. Ε, είναι στόχος που θέτει η συνθήκη στο άρθρο 174 ούτω ή άλλω. Αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε τους στόχους της συνοχή και βάσει της νομικής, ε, των νομικών προδιαγραφών που υπάρχουν. Έχουμε δει να υπάρχουν ε, εντάσεις μεταξύ των επιδόσεων, των τάσεων απλούστευσης, της αναθεώρησης της οικονομικής δικυβέρνησης. Βλέπουμε ε, οι εξελίξεις των τελευταίων 30 χρόνων να έχουν οδηγήσει σε μια διαφορετική διαστρωμάτωση των κανόνων με περισσότερη προβολή των αποτελεσμάτων που πρέπει να είναι γνωστά και στο κοινό. Όμως αυτό είχε κόστος και διοικητικό και στην καλή φήμη της πολιτικής συνοχής. Δυστυχώς μεταξύ των ενδιαφερομένων υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τις πρόσθετες υποχρεώσεις που βαραίνουν πλέον, πλέον τις αρχές διαχείρισης και τους δικαιούχους. Στο νέο περίοδο λοιπόν προγραμματισμού, η σύστασή μα είναι να επιδιώξουμε πραγματική απλούστευση. Πολλέ προσπάθειε απλούστευση έγιναν με βάση παλιότερε προτάσει, αλλά πρέπει να γίνουν ε, σοβαρές αλλαγές σε, πολλές, σε πολλούς τομείς της πολιτικής, όπου χρειάζεται βεβαίως. Η επιπλέον απλούστευση είναι σαφώ στόχος για τους δικαιούχους, αλλά ακόμα και για τι αρχές διαχείρισης, καθώς και τους αρμόδιους φορείς, που είναι διαρκώς αποσχολημένε σε διαδικασίε μεταρρύθμιση. Τελευταίο θέμα είναι η συμμετοχή των πολιτών και το πώ προβάλλεται η πολιτική συνοχή, πώς ε, διαφημίζεται. Είναι ένα σημαντικό θέμα και ειδικά στο σημερινό τοπίο με τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα να βρίσκονται σε έξαρση σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις προσπάθειες ε, ενημερωτικών εκστρατιών, προβολής και με τον στόχο 5, με, την, με το σύνθημα Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες πρέπει να προχωρήσουμε και στην Επιτροπή σας έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Μάλιστα εκπονούμε μια μελέτη που σύντομα θα ολοκληρωθεί για το πώς λειτουργούν τα μέσα μαζική ενημέρωση και επηρεάζουν αυτή την πολιτική στα διάφορα κράτη-μέλη. Βασική σύσταση σε αυτό το τομέα είναι να γίνει μια από τι πρώτε προτεραιότητε ε, το θέμα τη προβολή και τη επικοινωνία με δημιουργικέ λύσει. Το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ένας ε, πρωταθλητής της ε, προσέγγισης που να ε, απευθύνεται στους πολίτες. Δημοκρατικές καινοτόμες λύσεις, συμμετοχικός προγραμματισμός του προπολογισμού, αποφάσεις και συζητήσεις με εξεταστικές επιτροπές, με δημοσκοπήσεις, με διαβουλεύσεις και συμμετοχή και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό θα μπορούσε στη βιώσιμη ανάπτυξη με πιλωτικέ προσπάθειες να προχωρήσει στο μέλλον. Πάντω πρέπει να προσφερθεί ευκαιρία να συσφίξουμε του δεσμού με του πολίτε. Η Ευρώπη πραγματικά να έρθει πιο κοντά στου πολίτε και η αρχή τη ενεταιρικής σχέση που ήταν πολύ καινοτόμα για τη δεκαετία του 80 και του 90 να οδηγήσει σε ένα νέο εργαλείο διακυβέρνηση που να επιτρέψει να συσφίξουμε του δεσμού με του πολίτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Έχετε ερωτήσεις. Σημειώνω αυτούς που θέλουν να πάρουν το λόγο. Μάλιστα, κύριε Σπένικη. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να μιλήσω στα φιλανδικά, στη γλώσσα μου. Περιμένω λίγα δευτερόλεπτα να βάλετε τα ακουστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου έχει άμεση σχέση με την τελευταία παρουσίαση και την τελευταία πρόταση θα ήθελα να μιλήσω για την απλοποίηση, την απλούστευση και την μείωση της γραφειοκρατίας και του γραφειοκρατικού άχθους. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να έχουμε έναν πιο στρατηγικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή καθαρά στρατηγικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ξεκινάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στρεφόμαστε προς το κράτος μέλος, όπου οι περιφέρειες και οι διάφορες ε, περιφερειακές δομές πρέπει να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν. Αυτό πάντα σε συνδυασμό με το κράτος μέλος, με τις εθνικές αρχές και με την Ευρώπη τελικά, με την Επιτροπή. Καταλαβαίνετε όλο αυτό αποτελεί μια πολύ βαριά γραφειοκρατική διαδικασία η οποία ε, έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και μπορεί τελικά η οικονομία να είναι 20 ευρώ και όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία που βαραίνει όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις περιφερειακές αρχές θα πρέπει πραγματικά και οι περιφέρειες και οι δήμοι και οι κοινότητες και οι εθνικές αρχές αλλά και οι κομισιόν να συνεργαστούν έτσι ώστε αυτή η βαριά γραφειοκρατία να εξαλειφθεί. Πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλα παραδείγματα που θα δείχνουν ότι δεν έχουμε μειώσει ακόμα αρκετά την γραφειοκρατία. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σόπολ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και αναλύσεις σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον όσον αφορά τον πολλαπλασιαστή. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δημιουργούμε υποδομές, χτίζουμε υποδομές, οι οποίες όμως τελικά δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο ούτε στο επίπεδο ζωής, ούτε στην οικονομία των περιφερειών. Και αναφερθήκατε πολύ συγκεκριμένα στο τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με καλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, μιλήσαμε για βιωσιμότητα αυτών των πολιτικών. Χρειαζόμαστε όμως πραγματικές προτάσεις για να μετρήσουμε αυτήν την βιωσιμότητα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε από την αρχή του σχεδιασμού των έργων αυτών. Των έργων αυτών που τελικά θα καλούνται να διαχειριστούν και να λειτουργήσουν οι περιφερειακές αρχές. Μιλήσατε για εμπόδια. Μπορείτε να μου, που, να μου πείτε το ποσοστό των εμποδίων αυτών που προέρχονται από την Ευρώπη ποιο είναι σε σχέση με τα εμπόδια των εθνικών αρχών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια, όπως παραδείγματος χάρη είναι η διαφθορά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πείτε μου λοιπόν, τι επιβάλλει η Ευρώπη σε γραφειοκρατία, σε εμπόδια και τι επιβάλλουν τελικά τα εθνικά κράτη και οι περιφέρειες. Μιλήσατε επίσης για συνέργεια, για καλύτερη συνεργασία και είναι ενδιαφέρον να δούμε παραδείγματος χάρη τι κάνει η πολιτική συνοχή σε σχέση με άλλα προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες όπως το Horizon και άλλα. Έχετε εξετάσει τις πιθανές περαιτέρω συνέργειες. Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν απλούστερες διαδικασίες αλλού σε σχέση με αυτές που βλέπουμε όσον αφορά την εφαρμογή και την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Έχετε λοιπόν εξετάσει αυτές τις πιθανές συνέργειες, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστώ, Ολμπράιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Καταρχήν, Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική παρουσίαση που μας κάνατε. Αυτά τα δύο κέντρα έχουν εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες. Θα τους κάνω λοιπόν μια πολιτική ερώτηση. Πρόκειται για μια ανάλυση η οποία δεν έγινε για το Συμβούλιο ούτε για την Επιτροπή. Απευθύνεται σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή Ρέτζι τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ένα μεγάλο τμήμα της παρουσίασης των παρουσιάσεων έχω την εντύπωση ότι έχει γραφτεί με έναν αρκετά ολοκληρωμένο και γενικό τρόπο. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτά που μας παρουσιάσατε ισχύουν όποια και να είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα έχουμε μία προσέγγιση και μία τοποθέτηση της σημερινής Επιτροπής. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως εμάς σαν Επιτροπή Ρέτζη σήμερα είναι πώς θα πρέπει να τοποθετηθούμε, να αντιδράσουμε σε σχέση με την σαφή θέση της Επιτροπής. Όταν δηλαδή ξεκινήσει η συναπόφαση και όταν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Από τη μία είναι το θέμα της χρηματοδότησης για τις ε, περιφέρειες, για την Ήπεθρο και δεύτερον διάβασα πολύ προσεκτικά τις συστάσεις που μας προτείνατε όσον αφορά την επανενσωμάτωση στην περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Τι περιμένετε λοιπόν συγκεκριμένα από μας, εμείς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του τελικού κειμένου του κανονισμού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είστε εμπειρογνώμονες, γιατί κάποια πράγματα δεν τα βλέπω στην παρουσίασή σας. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει τη φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής, αλλάζει τους δίκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει να αλλάξουμε και τα κονδύλια για τη συνοχή. Μας ζητάει να αλλάξουμε τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των περιφερειών. Μα αλλάζει η πολιτική συνοχής. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή σας. Αλλάζει η έννοια της πολιτικής συνοχής για τα επόμενα χρόνια. Και συμφωνώ απολύτως με το θέμα της συνοχής των κονδυλίων και της χρηματοδότησης. Εσείς όμως, τι προτείνετε σε μας στην Επιτροπή Ρέτζη να συμφωνήσουμε ναι ή όχι με τις ε, πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Η Ρόζα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να προτείνω, κοιτάζοντα το πρώτο σημείο και την έλλειψη στρατηγικού πλαισίου για την πολιτική συνοχή που προκύπτει τη μελέτη. Δεν είναι μια λύση να φροντίσουμε να ταυτιστούν οι περίοδοι των κοινοβουλευτικών θητιών με την περίοδο προγραμματισμού, διότι τώρα απλώς πρόλαβα να κάνω μια πρώτη Μάλλον προλάβαμε να έχουμε μια πρώτη ανάγνωση όλων αυτών των ε, κειμένων και πολλοί συντονιστέ έχουν καταφέρει στου τριμμένου διαλόγου να προχωρήσουν τη δουλειά του. Όμω έχουμε διαφορετικά κείμενα με διαφορετικού προγραμματισμού στι διάφορε επιτροπέ. Και στην πολιτική συνοχή, λοιπόν, κλαθούν οι περιόδοι προγραμματισμού να συμπίπτουν με τι κοινοβουλευτικέ θητείε. Επίση, για την οικονομική διάσταση, την οικονομική διακυβέρνηση. Τι εννοείται ακριβώ με, την προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στι περιοχές, στους τόπους. Διότι αυτή η εδαφική προσέγγιση αφορά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εάν αυτό εννοεί, ε, μας απασχολεί πολύ εάν θα λάβουν κοινοτική διάσταση. Μπορούμε να το εξηγήσουμε καλύτερα, δηλαδή να εξηγήσετε εσείς οι υπεύθυνοι τη μελέτη, τι εννοείται με την εδαφική προσέγγιση και για την απλούστευση. Βεβαίω και το Κοινοβούλιο παροτρύνει σε περισσότερη απλούστευση. Ήθελα όμω να μου πείτε, παρόλο που συμφωνώ ότι τα ελλείμματα σε επίπεδο ε, αρχών τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικών φορέων έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι που να μπορούν να προγραμματίσουν ε, γρήγορα και να επιτρέψουν τη συμμετοχή σε σχετικές δημόσιες προμήθειες. Και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, για την καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Σίγουρα συμφωνούμε, διότι δεν είναι θέμα προπαγάνδας, καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική πρέπει να υπάρξει, αλλά θα πρέπει εγκαίρως και να ενημερώνει και για θέματα κρίσιμης σημασίας, όπως την λήξη προθεσμίας για συμμετοχή σε δημόσιους Καλό θα ήταν να επιβληθεί μάλιστα αυτό, αυτό και να περιλαμβάνει και την ενημέρωση για τα ταμεία της συνοχής και τα διαστατικά. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ με μια πολύ θετική αποτίμηση για τη μελέτη αυτή. Ε, πολλά σημαντικά στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν για μας ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και για την τωρινή μα συζήτηση και για τον ρόλο που επιθυμεί να αναλάβει η Επιτροπή μα και γενικότερα το Κοινοβούλιο. Σε σχέση με, το, με τη δομή της ομιλίας που ακούσαμε, με τα έξι σημεία, <clears throat> για την συνοχή που χρειάζεται τον καλύτερο συντονισμό των ε, κονδυλίων για την πολιτική συνοχή. Αυτό απαιτεί μεταρρυθμίσει και από πλευρά των κρατών. Πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τα κομβικά σημεία της πολιτικής συνοχής για να δούμε πώς θα ορίσουμε τις διάφορες εταιρικέ σχέσεις. Αυτό για την ώρα το συζητούμε με αφορμή τους σχετικούς κανονισμούς. Σαφώς συμφωνώ για την συνοχή των κονδυλίων λοιπόν, για το θέμα του Ταμείου για την, για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Βεβαίως η συνοχή εδώ έχει κρίσιμη σημασία να διαδραματίσει και επίσης είναι σημαντικό να ασχοληθούμε και εδώ με το θέμα της εταιρική σχέσης. Όμως, έχω εδώ μια διαφορετική άποψη. Το θέμα της εταιρική σχέσης και της ενίσχυση του τι είναι εταιρική σχέση θα μπορούσε να είναι θετικό, προσοχή όμως, στους κινδύνους που μπορεί να ελοχεύουν. Μπορεί να αυξηθεί το γραφειοκρατικό άχθος από ότι να μειωθεί. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε εδώ ιδιαίτερη προσοχή. Και η οικονομική διακυβέρνηση είναι σημαντική και βάσει των διαφορετικών κατευθύνσεων που ακολουθούν τη διαφορά κάτι μέλη. Για τη δίκαιη συμβιβαστική λύση που πρέπει να βρούμε μεταξύ του κεντρικού χαρακτήρα, τη κεντρική διοργάνωση και της εδαφικοποίηση, τέλος πάντων της ε, εξέτασης σε εδαφικό επίπεδο των διαφορών ε, προτάσεων και προγραμμάτων. Ένα πολύ σημαντικό σημείο και επ' αυτού νομίζω πρέπει να, να, να κάνουμε περισσότερη δουλειά και να το προσέξουμε ιδιαίτερα, τη συμμετοχή των πολιτών και την επικοινωνιακή πολιτική. Είναι σημαντικό να υπάρξει απλούστευση για να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας εδώ. Να αναλάβουν περισσότερα τα κρατη και να ορίσουν συστήματα απλούστερα. Διότι κάποιες φορές στην πράξη τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα από ό,τι θεωρητικά προβλέπονταν από τους όρους ενός προγράμματος, οπότε αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα και αυξάνει τις δαπάνες. Εάν το ψάχναμε λοιπόν σωστά, θα βλέπαμε τι δυσκολίες, τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ του τι ισχύει στις καλές πρακτικές που συχνά προβάλλονται και το τι γίνεται με μια περίπλοκη πραγματικότητα. Ευχαριστούμε κυρία Ντονάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα απλώς να προσθέσω εντάχει κάποιες δικές μου παρατηρήσεις για μερικέ μερικές πτυχές. Πρώτα απ' όλα για την οικονομική διακυβέρνηση. Καθόσον η αναφορά στην αιρεσιμότητα και τις περιφερειακές πτυχές είναι κρίσιμη σημασίας, παρόλα αυτά έχουμε και κάποιους συνδυασμού. Είδαμε τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν και τι πολιτικές ε, επιπλοκές στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στα κάτι μέλη. Το πώς ε, ταμιεύονται τα κονδύλια και πώς εκτελούνται, να υπόκειται σε όρους ε, που απαιτούν διαθεωτικές μεταρρυθμίσεις, ξέρουμε τι σημαίνει. Πολύ συχνά σημαίνει μεταρρύθμιση των εργασιακών πολιτικών, των πολιτικών για τις συντάξεις, οι ε, άλλες πτυχές, πολύ συγκεκριμένες της ε, εθνικής πολιτικής για την οικονομία. Αυτά προφανώς δικαίως ε, προσκρούν σε αντίσταση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν συμμερίζονται τις μεταρρυθμίσεις που εικάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι απαραίτητες αντιστέκονται οι κυβερνήσεις και πολλές φορές έχουν δείξει ότι δεν είναι και αποτελεσματικές θετικές στην ε, υλοποίησή τους, στην πράξη. Η αιρεσιμότητα λοιπόν αυτή, το σύστημα υποβολής σε όρους, που απαιτεί η ευρωπαϊκή πολιτική από τις ε, δυσκολία χώρες, τώρα και με το σύστημα των κονδυλίων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους τριγμούς και προβλήματα χρειάζεται περισσότερη δημοκρατική εμπλοκή των πολιτών. Διότι εάν αφήναμε στου πολίτε των μελών το δικαίωμα να εκφράσουν τη δική του γνώμη για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι πολλοί θα ε, διαφωνούσαν. Το σύστημα των ευρωπαϊκών κονδυλίων βασίζεται στην ε, υπόθεση ότι όλοι συμβάλλουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό με μεγάλα ποσά. Η Ιταλία είναι από τους βασικούς ε, συμβάλλοντες μεταξύ των 100 μελών. Άρα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά μια αποπληρωμή των όσων έχουν ήδη δοθεί ε, από το κάτω μέλος αρχικά για να καταρτήσει ο ευρωπαϊκός προπολογισμός. Εάν τώρα εδώ επιβάλλονται και κριτήρια, όροι και ρεσιμότητε, με πολιτικέ ενδεχομένω σκοπιμότητε, πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό κίνδυνο από πλευρά των πολιτών αυτό θα γίνει αντιληπτό ω ε, άδικο και μη ε, σωστό. Το σύστημα των ευρωπαϊκών κονδυλίων λοιπόν και το όφελος μέσω της πολιτικής συνοχής για τις ε, περιοχές, τις, τις περιφέρειες της Ευρώπης είναι σημαντικό. Αλλιώς μπορεί να το θέσουμε σε κίνδυνο. Καλό θα ήταν να σκεφτούμε και να προσέξουμε το σύστημα αυτό της ερεσιμότητας Ενδεχομένως να πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις να πρέπει να επαναορίσουμε τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει, αλλά με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Και η τελευταία παρέμβαση από την κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι παρουσιάσεις αυτές που μόλις έγιναν ουσιαστικά μου δημιουργούν ε, ανάμεικτα συναισθήματα και από τη μία Αντικατοπτρίζεται αυτά που θα πρέπει να είχαμε κάνει πριν όμως μας έρθει και εξετάσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Σήμερα όμως έχουμε λάβει την πρόταση της Επιτροπής, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής των τροπολογιών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Και η ερώτηση που επαναλαμβάνουμε όσον αφορά την αιρεσιμότητα έχει απαντηθεί από εμάς. Την απόφαση μας την έχουμε λάβει. Δεν θέλουμε μακροοικονομικές προϋποθέσεις και όρους. Και βεβαίως, ποια είναι η στήριξη των κρατών μελών Ίσως κάποια από αυτά τα μακροοικονομικά κριτήρια και όρους να στηριχθούν από κάποια κράτη-μέλη. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι είναι κάτι θετικό, αλλού όμως ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για την στρατηγική που θα επιλέξουμε και που θα επιλέξουν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα την συνοχή, την εδαφική συνοχή, ξέρετε ότι πόσο θα υποχωρήσουμε όσον αφορά άλλου είδους κεντρικά προγράμματα, άλλου είδους ευρωπαϊκές αποφάσεις, το... Η χρηματοδότηση μέσω του Γεωργικού Ταμείου έχει ήδη αποφασιστεί και φυσικά δεν νομίζω ότι πρέπει να μας πείσετε όσον αφορά τον κανονισμό αυτό και αν θα είναι κανονισμός πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα πάντα. Εδώ και μισό χρόνο περίπου, ένα εξάμεινο συζητάμε το θέμα αυτό. Θα έπρεπε τότε να μας είχατε πείσει. Σήμερα είμαστε εδώ μπροστά σε νέους συναδέλφους, οι οποίοι ναι μεν πρέπει να ενημερωθούν, αλλά ουσιαστικά κάνετε σαν να μην είχαμε πάρει θέση. Αυτή η παρουσίαση για μένα ε, είναι μια παρουσίαση που μου δημιουργεί πάρα πολύ ανάμεικτα συναισθήματα και δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των ομιλητών και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπόγκοβιτς ε, που είναι πραγματικά ο τελευταίος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας για την παρουσίαση της μελέτης που θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας. Έγινε μια πολύ καλή επισκόπηση της πολιτικής συνοχής στη μελέτη, αλλά συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν για το ρόλο της δικής μας Επιτροπής. Και στο νέο απολυτής δημοσιονομικό πλαίσιο συμφωνούμε όλοι ότι η γραφειοκρατία είναι μείζον πρόβλημα της πολιτικής συνοχής. Επίσης, ανάλογα με τη χώρα και την περιφέρεια, δεν είναι όλο το προσωπικό που ασχολείται με την πολιτική συνοχή κατάλληλα ενημερωμένο. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ο πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Συνοχής είναι να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το έχω επισημάνει πολλά και στο παρελθόν. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε με την αστιφιλία, με την έξοδο από την Ήπεθρο, με υπερφόρτωση των ε, μεγάλων αστικών κέντρων ή συγκέντρωση πληθυσμιακή σε, σε μερικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε την κατανομή των κονδυλίων. Μερικά κονδύλια δεν έφτασαν στις χώρες της συνοχής και διαπιστώνουμε και επίσπευση κάποιων αρνητικών τάσεων αντί για ε, αναστολή τους. Υπάρχει το 4,4, αλλά ε, στη σελίδα 25 έχουμε την βουλή για τα έξυπνα χωριά, είμαι υπέρ. Στο κεφάλαιο 5 μιλούμε για την ανοιχτή διάσταση της πολιτικής συνοχής. Τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πολλά στο αστικό θεματολόγιο, αλλά όχι αρκετά στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στα έξυπνα χωριά για παράδειγμα. Ελπίζω λοιπόν στους επόμενους μήνες να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας και στο θέμα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ήπεθρο και να δούμε πόσα κονδύλια θα διατεθούν για να υλοποιήσουμε τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής συνοχής και να αποτρέψουμε την ερήμωση της υπαίθρου. Δεν θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την αστιφιλία και να έχουμε συσσόρευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μόνο στα αστικά κέντρα ή περισσότερο στη Δυτική Ευρώπη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Καλή πολιτική συνοχής λοιπόν και δεν θα πρέπει να είναι συνέπεια της πολιτικής συνοχής η απερίμωση της υπαίθρου, θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην διαφύλαξη του πληθυσμιακού δυναμικού και των αγροτικών περιοχών και της υπαίθρου. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, τώρα όντως ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Η συζήτηση ήταν πολύ πλούσια και η μελέτη σας έγινε πολλά ζητήματα και απορίες και θέτει κάποια βασικά ερωτήματα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίθετα με τον συνάδελφο Όλμπριχτ, εγώ θεωρώ ότι όντως ρισκάρατε και πήρατε κάποιες αποστάσεις από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό πραγματικά είναι ρίσκο. Πάντως ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Ρέγκη Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, έχει ήδη λάβει θέση για τα ερωτήματα που εντοπίσατε και η θέση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αυτή που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ε, η διαπραγματευτική εντολή που θα είναι ο μύτος Αριάδνης για μας και για τις ε, μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αναφερθήκατε και στο ζήτημα της εταιρική σχέσης. Και αυτό το θέμα το εντοπίσαμε στην Επιτροπή μας και θα είναι από τα βασικά στοιχεία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Και σε αυτό το σημείο θα σταθούμε και θα το υποστηρίξουμε. Αναφερθήκατε και σε μία ανησυχία σας σε σχέση με το διαχωρισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης από την υπόλοιπα ταμεία ε, του, του ΕΦΣΙ, του ΕΤΣΕ, Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Εμείς είμαστε κατά επίσης. Ε, πολύ άριθμα είναι τα ζητήματα που εγείρατε και καταλήξαμε σε πολλά κοινά συμπεράσματα. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής λαμβάνει χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια περίπλοκη κατάσταση. Και όπως ε, αναφέρετε και εσείς ακροθυγός στην μελέτη σας, η πολιτική συνοχής δημιουργήθηκε και έγινε θύμα άδικων επιθέσεων. Γιατί υπάρχει, όπως επισημαίνετε και εσείς, ένα πρόβλημα συνέπειας μεταξύ των διαφόρων ταμείων και συνοχής μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Και δυστυχώς ε, δεν ε, εστερνίζονται όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους στόχους που κατοχυρώνει το άρθρο 175 της Συνθήκης. Και θα ήθελα να επιθυμίσω ότι οι στόχοι της συνοχής θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις πολιτικές. Η δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για σας και θα σας δώσω μετά το χρόνο να απαντήσετε. Μιλήσατε για την ανάγκη να εμπλέξουμε τους πολίτες, να κινήσουμε το ενδιαφέρον τους και να έχουμε σε κάποιες προτάσεις ε, ευρηματικής δημοκρατικής εφαρμογής. Έχετε πιο συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε πιο ενεργά τους πολίτες στην διαδικασία αυτή. Πάντως, τα θεμελιώδη προβλήματα που εντοπίζει η μελέτη σας και που είχαμε ζητήσει στις αρχές του χρόνου, ε, βέβαια μεσολάβησαν οι εκλογές και ακριβώς το γεγονός ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο κοινοβουλευτικές θητείες οδήγησε κάποια καθυστέρηση. Πάντως ε, συμφωνούμε ε, με τα προβλήματα που επισημάνατε. Και σίγουρα οι προτάσεις θα μας εμπνεύσουν στο μελλοντικό μας έργο. Και έχετε τώρα εσείς το λόγο για να απαντήσετε στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος της μελέτης, να προκαλέσει ζωηρές ε, συζητήσεις ε, και σχόλια και από εσά για την παρούσα κατάσταση και το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Θα κάνουμε μια επισκόπηση των βασικών θεμάτων, μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την παρουσίαση απόψεων διαφόρων ε, ενδιαφερομένων για την πολιτική και προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε μέσα σε 40 σελίδες για να κατατοπίσουμε κυρίως τα νέα μέλη της Επιτροπής ΡΕΓΚΙ για να έχουν κάποια σημεία αναφοράς με βάση τη μελέτη μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία που επισημάνατε και εσείς πρόεδρε και ο κύριος Γιάνν Όλμπριχτ, σίγουρα θα πρέπει να εμείνει στα ναρά απόψη η Επιτροπή ΡΕΓΚΙ να υπερασπίσει τις αρχές που ανέκαθεν υποστήριζε τα θέματα της εταιρικής σχέσης, της πρόθεσης, της ανάπτυξης των πόλεων, τη διαφύλαξη της συνοχής, του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής και αύξηση της προσθέμενης αξίας της πολιτικής, όπως είπε και η Φραντσέσκα Ντονάτο. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων να αναδείξουν την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής και στις εσωτερικές πολιτικές. Επίσης αναφερθήκατε πολύ σε απλούστευση και στη στρατηγική προσέγγιση. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συνέργειες και η συνέργεια της πολιτικής συνοχής με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί σε πολλά άρτια στρατηγικά σχέδια για μια συνεκτική προσέγγιση στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε μια τέτοια συνοχή. Ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τη χρηματοδότηση διαφόρων πολιτικών. Και έχουμε, είχαμε στο παρελθόν πριν από μερικά χρόνια εκπονήσει σχετική μελέτη, στην οποία σα παραπέμπω ενδιαφέρεστε. Δεν αναλύσαμε ε, λεπτομεριακά τα θέματα των πολλαπλασιαστικών ε, αποτελεσμάτων στην οικονομία, το κόστος της ε, αηφορίας. Όλα αυτά όμως υπάρχουν στη στοσέλη της Επιτροπής ε, και υπάρχουν πολλές μελέτες που ποσοτικοποιούν αυτά τα επιμέρους ζητήματα. Το θέμα του κανονιστικού υπερθεματισμού, του gold plating, είναι πρόβλημα όταν οι εθνικές αρμόδιες αρχές προσθέτουν ε, στρώματα νομοθετικά. Αλλά δεν είναι μόνο θέματα κανονιστικού υπερθεματισμού. Είναι και αιτήματα από τις ε, αρμόδιες αρχές για διευκρινήσεις κάποιων αφήσιμων άρθρων ή κάποιων διατάξεων που χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας και διευκρίνησης. Και όλα αυτά ενισχύουν το γραφειοκρατικό άχθος και το γραφειοκρατικό κόστος. Αναφέρθηκε, κα... από κάποιον ότι οι πολίτες, το χώρο που είναι καθαρή συνεισφορής, δεν βλέπουν την αξία μιας τέτοιας προσέγγισης. Μάλιστα, συναντήσαμε 250 πολίτες από 17 περιφέρειες και αυτό διαπιστώσαμε ότι οι πολίτες θέλουν να έχουν λόγο στη χρηματοδότηση της πολιτικής. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακέ οι γνώσεις τους ε, για τις χρηματοδοτήσεις κάποιων προγραμμάτων και θέλουν ε, μια πιο κεντρική ε, προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και να έχουν λόγο στη διαμόρφωση χρηματοδότησης αλλά φαίνεται ότι επικοινωνιακά δεν έχει φτάσει στους πολίτες το πλεονέκτημα της πολιτικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μας, όντως θα μπορούσατε να μας προσάψετε κάποια αργοπορία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, γιατί η δημοκρατία δεν σταματά πουθενά, ούτε το νομοπαρασκευαστικό έργο. Οπότε οι στάσει ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εφαρμογή και μελλοντικέ μεταρρυθμίσει. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε και το ιστορικό της πολιτικής και ε, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να παρουσιάσουμε την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως φαίνεται από τις διάφορες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις του. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Πολλοί ρώτησαν τι θα πει εδαφικοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης, η περίληψη της εδαφικής προσέγγισης δηλαδή. Στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα ε, διαπιστώνουμε ότι αυτές δεν προσαρμόζονται στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το ρόλο έχει ο προγραμματισμός των προγραμμάτων και των εταιρικών σχέσεων. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση, αλλά θα πρέπει να να το αναγνωρίσουμε αυτό και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, σε ένα πιο στρατηγικό επίπεδο. Γιατί όταν φτάνουμε στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή δεν είναι ε, σαφές ότι θα εφαρμοστεί στις διαπραγματεύσεις η εδαφική προσέγγιση της οικονομικής διακυβέρνηση. Κάποιες περιφέρειες και κάποιες χώρε είναι επικριτικές ε, ε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και πολύ φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο ε, θα αναδείξει τις διαφορές ε, μεταξύ των περιφερειών. Θα πρέπει όμως να γίνει αυτή η συζήτηση και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να ε, εξορροπήσουμε αυτές τις διαφορές. Σε ό,τι αφορά την ανάμειξη των πολιτών, την εμπλοκή των πολιτών και το σχέδιο αυτό, ε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πιο λεπτομεριακά σαφή παραδείγματα. Αλλά πιστεύω ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοια παραδείγματα δημοκρατικής καινοτομίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πολλές ε, μορφές ε, δημοκρατικού διαλόγου με τους πολίτες. Και πρόκειται για μια νέα προσέγγιση που τη βλέπουμε ήδη. Στη Σκωτία, για παράδειγμα, όπου διαμένω, ε, υπάρχει ένα ταμείο για την συμμετοχική χρηματοδότηση. Και έχουμε πολλά παραδείγματα σε άλλες πολιτικές. Όχι όμω την πολιτική συνοχή. Κακώ, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, πιο ενεργό συμμετοχή και των πολιτών στην πολιτική συνοχή. Γιατί πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε τους πολίτες ε, να αναμειχθούν στην εφαρμογή αν τους έχουμε αγνοήσει στο προηγούμενο ε, επίπεδο, το επίπεδο της χάραξης και της διαμόρφωσης της πολιτικής συνοχής. Αυτά προ τα βασικά σημεία και αν ξέχασα κάτι, πολύ ευχαρίστω να επανέλθω αργότερα. Merci beaucoup pour vos réponses. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της ανάλυσης της μελέτης σας και πραγματικά όταν τη διάβασα μου επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ορθή θέση τη θέση που εξάλλου θα υπερασπιστούμε και θα προωθήσουμε και στον τριμερή διάλογο. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ένα σημαντικό σημείο, διότι θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μάρκ Λεμέτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε τέτοιου είδους ε, ανταλλαγές απόψεων είτε με τον ίδιο τον ή την Επίτροπο είτε με τον Γενικό Διευθυντή της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Λεμέτρα είναι διοικητικός, δεν είναι πολιτικός και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε να του κάνουμε, άλλες θα απευθύνουμε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στον ή υποψήφιο επίτροπο για περιφερειακά θέματα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Λεμέτρη είναι εδώ για να μας παρουσιάσει την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων, την χρήση των κονδυλίων την παρακολούθηση της περιφερειακής πολιτικής από την Γενική του Διεύθυνση. Έχετε το λόγο και με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα πολύ προστατευτικά σας λόγια και ελπίζω να έχουν αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι εκ νέου εδώ προσκεκλημένος από την Επιτροπή Ρέτζι. Θυμάμαι την τελευταία μου ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή σας με το ένα δέκατο συμμετοχή από αυτή που βλέπω εδώ και ελπίζω πραγματικά ότι θα συνεχίσετε αυτήν την επιμέλεια και την επιμελή παρουσία σας εδώ έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω όλους ε, για την εκλογή σας, τα νέα μέλη. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω που επιλέξατε αυτήν την Επιτροπή. Ελπίζω ότι η συμμετοχή σας στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για μια Επιτροπή που τα επόμενα χρόνια και σίγουρα τους επόμενους 12 ε, μήνες ε, θα ασχοληθεί με στρατηγική σημασία υποθέσεις. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε για την εκλογή σας, καθώς και τους αντιπροέδρους της Επιτροπής. Σας συγχαίρω για την ε, πολύ συγκεκριμένη εκλογή σας και φυσικά θα ήθελα να αναφερθώ και στην Επίτροπο Κρέτσου με την οποία είχα τα τελευταία τρία χρόνια εξαιρετική συνεργασία για θέματα πολιτικής συνοχής. Είμαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα να έρθω εδώ νωρίς στο ξεκίνημα των εργασιών της Επιτροπής σας, διότι πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά επίγοντα η μετάβαση από τη μία θητεία στην άλλη δεν θα πρέπει να μας καθυστερήσει. Χρειάζεται εδώ έγκαιρη λήψη αποφάσεων για θέματα δημοσιονομικά και για θέματα μέλλοντος και προοπτικών της πολιτικής συνοχής. Φυσικά και είμαστε στη διάθεσή σας. Υπάρχουν εδώ πολλά νέα μέλη. Νέα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νέα μέλη εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και πιστεύω ότι η ιστορία της περιφερειακής πολιτικής, τα μέχρι τώρα γεγονότα αλλά και οι προοπτικές για το μέλλον είναι κάτι που σας έχει παρουσιαστεί. Εγώ δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα αναφερθώ κυρίως σε τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι μια ενημέρωση για σας όσον αφορά τους τελευταίους μήνες και την πολύ συγκεκριμένη υλοποίηση της προγραμματικής περίοδου 14-20, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Το δεύτερο θέμα που θα θίξω είναι ποια είναι τα πρακτικά βήματα όσον αφορά την προετοιμασία της επόμενης περίοδου, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και το τρίτο και σημαντικό σημείο θα είναι το να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις καθοριστικές πτυχές του οράματός μας για την ε, πολιτική της συνοχής για τα επόμενα δέκα χρόνια. Έχω και κάποιες διαφάνειες, τις οποίες βλέπετε στην οθόνη. Εγώ δεν τη βλέπω την παρουσίαση, ελπίζω εσείς να την βλέπετε καλύτερα από μένα. Θα ήθελα καταρχήν σε αυτή τη διαφάνεια να σας υπενθυμίσω τη συμμαχία, τη σημασία, συγγνώμη, της πολιτικής συνοχής σε σχέση με τον ε, προϋπολογισμό. Βλέπετε ότι είναι περίπου το 1 τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το 14 με 75 εκατομμύρια το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με 97 δισεκατομμύρια. Βλέπετε τη σημασία των τριών αυτών τρόπων χρηματοδότησης και βλέπετε και τι αντιστοιχεί σε εμά στη δική μας Γενική Διεύθυνση και τι αντιστοιχεί στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Η περίοδος 14-20 χαρακτηρίζεται και από μια σημαντική καινοτομία. Συγκεκριμένοι δείκτες επιδόσεων έχουν αρχίσει να λειτουργούν, να εφαρμόζονται και θα γίνει ένας απολογισμός στο τέλος της περίοδου αυτής. Εδώ βλέπετε κάποια από τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία χρησιμοποιούμε αυτούς τους ποσοτικούς δείκτες. Και βεβαίως πολλά από αυτά έχουν άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες μας. Πρώτον, θέσεις απασχόλησης, βελτίωση υπηρεσιών που αφορούν την υγεία. 55 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης υποφελούνται σήμερα από πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας. καθώς και βελτιωμένη φροντίδα για τα παιδιά και στον τομέα της εκπαίδευσης, βελτιωμένες υποδομές για 6,9 εκατομμύρια παιδιά και σπουδαστές βελτιωμένη κατανάλωση ενέργειας για πάνω από 800.000 νοικοκυριά. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι στόχοι έχουν άμεσες θετικές επιπτώσεις στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς θα πετύχουμε και θα βελτιώσουμε την υλοποίηση αυτών των στόχων και αυτής της πολιτικής. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ικανοποιητική. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, τη βελτίωση όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 7-13, 2007-2013, μια περίοδο δηλαδή που χαρακτηρίζεται από μια σοβαρότατη κρίση. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα, δηλαδή 14-20, Το 2007-2013 είναι η πάνω γραμμή και η κάτω γραμμή αφορά την σημερινή περίοδο. Βλέπετε ότι οι δύο αυτές γραμμές δυστυχώς αποκλίνουν και η απόκλησή τους αυξάνεται. Είμαστε στο τέλος του έκτου έτους αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου και ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει ούτε το 1 τέταρτο των ποσών. Είδατε γιατί ποσά αναφερόμαστε. 380 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι εξαιρετικά μη ικανοποιητικό και καλούμεθα να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αυτά και τους ρυθμούς υλοποίησης το ταχύτερο δυνατόν. Το 2020 σας φαίνεται ότι θα είναι ένα πολύ καλό έτος. Όμως το μισό από η μισή από τους στόχους μας δεν θα έχουν υλοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά βλέπουμε ότι οι κανόνες για αυτή την περίοδο έχουν χαλαρώσει και επιτρέπουν από τα κράτη-μέλη να περάσουν στο N plus 3. Δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν για τρία περαιτέρω χρόνια τις δυνατότητες υλοποίησης. Γιατί η πολιτική συνοχή έχει γίνει τόσο δύσκολη, έχει πάψει να λειτουργεί, δεν νομίζω. Απλώς οι κανόνες είναι εξαιρετικά χαλαροί και αυτό επιτρέπει σε όλους, σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλα τα επίπεδα να αναβάλουν, να καθυστερούν και να χρονοτριβούν. Και αυτό γίνεται και εις βάρος της ποιότητας, αλλά και εις βάρος πραγματικά των επιπτώσεων, των θετικών επιπτώσεων στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα δεν βλέπουν το αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε πραγματικά την εφαρμογή και την υλοποίηση, αλλιώς και εμείς ουσιαστικά ενισχύουμε την ύφεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η δυνατότητα αντίδρασής μας είναι αυτή, αυτή που βλέπετε. Θα σας δείξω και μια άλλη πτυχή της ίδιας ιστορίας που είναι η επιλογή των σχεδίων και προγραμμάτων. Όσον αφορά την επιλογή, τα πράγματα έχουν παραμείνει σταθερά σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013. Αυτό βεβαίως δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από τα, τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτική συνοχή, γιατί η επιλογή των σχεδίων δεν σημαίνει τίποτα όσον αφορά την αλλαγή της καθημερινής ζωής των πολιτών μας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται μόνο στα χαρτιά. Αυτές οι δύο διαστάσεις λοιπόν, οι συγκεκριμένες δαπάνες από τη μία, η επιλογή των σχεδίων από την άλλη, παρουσιάζονται εδώ σε αυτό το διάγραμμα. Σας δείχνουμε δηλαδή τι ακριβώς κάνει το κάθε κράτος μέλος και πώς τοποθετείται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Βλέπετε λοιπόν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Όσο πιο ψηλά βρίσκεστε, τόσο πιο ε, πολλά προγράμματα έχετε υλοποίησει. Και εδώ βλέπετε και την γραμμή που οριοθετεί την επιλογή. Πόσα προγράμματα, πόσα σχέδια έχουν επιλεγεί και όπως σας είπα, λιγότερο από 25% αν βγάλετε τις προκαταβολές όσον αφορά τις πολύ συγκεκριμένες δαπάνες. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν που βρίσκονται δεξιά είναι μάλλον καλοί μαθητές όσον αφορά την υλοποίηση. Αντίθετα, οι χώρες που βρίσκονται αριστερά είναι πιο καθυστερημένες. Όσον αφορά τις πάνω χώρες και τις κάτω χώρες, αυτό αφορά την επιλογή των προγραμμάτων. Σε αυτήν την διαφάνεια αντικατοπτρίζουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις, την υλοποίηση που έχουμε συλλέξει καθημερινά από στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Πραγματικά, αν χρειάζεστε στοιχεία, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το πόσο έχουμε προχωρήσει στη δική σας χώρα, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία αυτά στο διαδίκτυο. Η βάση δεδομένων ονομάζεται Open Data Platform. Όπως σας έλεγα, μας αφορούν οι επιδόσεις και έχουμε στοχεύσει ιδιαίτερα στην περίοδο 14-20 στην μέτρηση των επιδόσεων. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο χρησιμοποιούμε με κίνητρα για συγκεκριμένες προτεραιότητες στο εσωτερικό των προγραμμάτων και σχεδίων. Ήθελα εδώ να αναφέρω ότι το 6% των διαθέσιμων ποσών κρατούνται στην αρχή του προγράμματος και στο τέλος του πέμπτου έτους, δηλαδή το 2018, θα απελευθερωθούν ή όχι τα ποσά αυτά από τη στιγμή που έχουν προχωρήσει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το 2018 δηλαδή κάναμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μία αξιολόγηση. Πρόκειται για κάτι σχετικά πρόσφατο και μπορώ να σας δώσω τα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης των επιδόσεων. Αυτό το 6% που είχαμε κρατήσει ουσιαστικά ανταποκρίνεται για όλα τα προγράμματα σε ένα ποσό που φτάνει τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 22 από αυτά τα 27, δηλαδή το 80% αυτού του ποσού, θα δοθεί στα αρχικά προγράμματα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή το 80% αυτού του ποσού θα δοθεί καθότι το 80% των στόχων έχει υλοποιηθεί. Αυτό είναι καλό, ικανοποιητικό σαν αποτέλεσμα. Αντίθετα, αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που απομένουν από τα 22 στα 27 θα πρέπει να δοθούν, θα μεταφερθούν σε προγράμματα που είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις και των οποίων οι προτεραιότητες υλοποιήθηκαν με τους ε, ρυθμούς όπως είχαν προκαθοριστεί. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή θα υπάρξει ένας νέος προγραμματισμός και έχω να κάνω και δύο σχόλια γι' αυτό που αφορά το μέλλον. Ποιες είναι οι προτάσεις μας για αυτή την κατάσταση. Πρώτον, θεωρούμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε αυτή την αξιολόγηση των επιδόσεων που για πρώτη φορά λειτουργεί. Δεύτερον, αυτή τελικά η αξιολόγηση όταν γίνει ο επαναπρογραμματισμός και ολοκληρωθεί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έχει κάποια απογοητευτικά αποτελέσματα ως ένα βαθμό. Γιατί? Διότι πρόκειται για κάτι το πολύ αυτόματο, μηχανικό. Δηλαδή βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε αν είμαστε κοντά στους στόχους, την υλοποίηση του στόχου και καμιά φορά ο στόχος από την αρχή έτσι όπως τοποθετήθηκε ίσως να ήταν πολύ φιλόδοξος ή πολύ συντηρητικός. Και τελικά θα βρεθούμε τελικά με κάποιες προτεραιότητες οι οποίες δεν θα στηριχθούν, θα μεταφερθούν κονδύλια σε κάποιες άλλες προτεραιότητες που αν είχαμε αρχικά την ε, δυνατότητα να επιλέξουμε, δεν θα το είχαμε κάνει ποτέ. Γι' αυτό και θα προτείνω κάτι άλλο για το μέλλον. Έναν πιο ποιοτικό μηχανισμό και όχι τόσο αυτόματο, έτσι ώστε τα, την δεύτερη χρονιά 5 συν 2 να μπορεί να γίνει μία ολοκληρωμένη ε, και πολιτική αξιολόγηση έτσι ώστε να δούμε με προσοχή τα τελευταία γεγονότα, το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν και υλοποιήθηκαν τα επιμέρους προγράμματα. Η εμπειρία μας λοιπόν με αυτήν την ε, αξιολόγηση των επιδόσεων, πώς θα μοιραστεί και θα κατανεμηθεί αυτό το αποθεματικό ποσό, τελικά μας έχει οδηγήσει στην πεποίθηση ότι θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον και να επεξεργαστούμε περαιτέρω την νέα μας πολιτική. Αυτά τα πέντε δις τελικά θα μεταφερθούν από τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία παρουσιάζουν περισσότερες αδυναμίες όσον αφορά την υλοποίηση. Αυτές οι αδυναμίες έχουν άμεση σχέση και με τους ρυθμούς υλοποίησης. Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, και Ρουμανία. Είναι οι τέσσερις χώρες αυτές από τις οποίες θα μεταφερθούν αυτά τα 5 δισεκατομμύρια. Η πολιτική συνοχής και στο παρελθόν πολλές φορές ήταν αντικείμενο επικρίσεων ότι δηλαδή δεν υπήρχε πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ότι υπάρχουν ποσά τα οποία εδώ και 20 χρόνια δεν είχαν απορροφηθεί κτλ για την περίοδο 2007-2013 έγινε πολύ εντυπωσιακή πρόοδος με επιτάχυνση των ρυθμών και σήμερα πρέπει να σας πω ότι μόνο 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παραμείνει λιγότερο δηλαδή από το 1% του συνολικού ποσού για το 2007-2013 δεν έχει πραγματικά δαπανηθεί. Αλλά θα υπογραμμίσω ότι το 2007-2013 δεν υπήρχε αυτό το νη συν 3, αλλά ήμασταν ακόμα στον προηγούμενο κανόνα νη συν 2. Δηλαδή η αναβολή μπορούσε να γίνει από τα κράτη-μέλη μόνο για δύο χρόνια και να ξοδευτεί το ποσό τα δύο επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά το 2021 27 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα και να προκαταλάβει τις αρχές που είναι αρμόδιες για να νομοθετήσουν, εσάς δηλαδή, αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Θέλουμε όμως να προετοιμάσουμε την περίοδο αυτή έτσι ώστε να υπάρξει μία υιοθέτηση των εκτελεστικών προγραμμάτων, των εταιρικών σχέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως, έτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου του 2021 να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η νέα προγραμματική περίοδος. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Όπως ξέρετε, προτείναμε να ενισχύσουμε τη διασύνδεση μεταξύ πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ε, οικονομικής διακυβέρνησης δηλαδή. Και το τελευταίο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του 2019, από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή έχουν επεξεργαστεί την ανάλυση της Επιτροπής, τα συμπεράσματα της Επιτροπής όσον αφορά δύο τομείς. Πρώτον, τις ε, διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών των κρατών μελών και τις επενδυτικές ανάγκες που όπως βλέπουμε θα οδηγήσουν σε νέες προτεραιότητες όσον αφορά την πολιτική συνοχή για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όλα αυτά ουσιαστικά έχουν υποβληθεί στις λεγόμενες εκθέσεις ε, για την κάθε χώρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και μάλιστα σας καλώ να ενημερωθείτε, να διαβάσετε την έκθεση για τη χώρα την οποία γνωρίζετε και σας αφορά άμεσα και στα παραρτήματα της κάθε έκθεσης για την κάθε χώρα παρουσιάζει βάση της ανάλυσης των στόχων τι θεωρεί προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θεωρούμε ότι η βάση της ανάλυσής μας θα πρέπει στην επόμενη προγραμματική περίοδο να θεωρηθεί προτεραιότητα. Και μάλιστα προτείναμε μια νέα αρχιτεκτονική για την πολιτική συνοχής. Θα επανέλθω σε αυτό με πέντε στόχους ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες έχουμε υπογραμμίσει σε αυτά τα παραρτήματα για τα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πάρω τις δύο ακραίες περιπτώσεις. Από τη μία πάνω-πάνω βρίσκεται κάποια κράτη-μέλη που έχουν θα έλεγα 10-15 ευρώ το έτος ανάτομα που είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία και το Λουξεμβούργο. Πρόκειται για χώρες οι οποίες στοχεύουν όσον αφορά τις δαπάνες στην πολιτική συνοχή σε δύο προτεραιότητες. Πρώτον, πιο έξυπνη Ευρώπη, δηλαδή καινοτομία, ανταγωνισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ιδιωτικοποίηση. Και τέσσερα, στόχος τέσσερα που είναι το ανθρώπινο δυναμικό βελτίωση των προσόντων, των δεξιοτήτων κτλ. κτλ. Στο άλλο άκρο, κάτω-κάτω δηλαδή, έχετε αρκετά κράτη-μέλη θα έλεγα, όπου υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στην πολιτική συνοχής. Και εδώ η πολιτική συνοχής μπορεί πραγματικά να στηρίξει επενδύσεις και δυνατότητες επενδύσεων. Δεν μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, το κλίμα, διασυνδέσεις ε, υποδομών, μεταφορές, θέματα διασύνδεσης ε, των δικτύων ενέργειας, ψηφιακή διασύνδεση και μια προσέγγιση που αφορά τον στόχο 5 για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Εμείς ήδη Έχουμε κάνει κάποια γεγονότα που αφορούν το κάθε κράτος μέλος για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και χαίρομαι γιατί αυτά πήγαν πολύ καλά, είχαμε πολύ επιτυχία και είναι ένα είδος κινήτρου αν θέλετε για τα κράτη-μέλη για να αρχίσουν να οραματίζονται την επόμενη προγραμματική περίοδο τι θα ήθελαν να επιλέξουν σαν δράσεις και ιδιαίτερα να αποδραματοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτόν τον ε, δεσμό μεταξύ Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, Πολιτικής Συνοχής, Περιφερειακής Πολιτικής, γιατί με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το είχαμε προωθήσει, για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να τους βοηθήσουμε να οραματιστούν, αν θέλετε, τις νέες τους προτεραιότητες για το μέλλον. Πολύ γρήγορα και για να εκμεταλλευτούμε αυτό το ρυθμό που ήδη υπάρχει, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να μας στείλουν κάποια προσωρινά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα μπορούσαν να δώσουν κάποια πρώτα προσωρινά σχέδια προγράμματος και προγράμματα υλοποίησης. Και πότε θα μπορούσαν να μας δώσουν τα τελικά προγράμματα που θα μπορούσε να εγκρίνει η Επιτροπή εν τέλει. Όλα τα κατημέλια απήντησαν. Και όλοι μας έδωσαν τέτοιες ενδείξεις που επέτρεψαν να ελπίζουμε, να ευελπιστούμε μάλλον ότι μπορούν να υιοθετηθούν προγράμματα στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή όλα να ξεκινήσουν ε, στη σωστή στιγμή. Βεβαίω όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το αν οι συνομοθέτε θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο. Αλλά πραγματικά ευελπιστούμε ότι με την διαθεσμική αλληλεπίδραση όλα θα πάνε καλά στο τέλος της επόμενης χρονιάς και θα υπάρξει συμφωνία στα επιμέρους νομικά κείμενα. Να στραφώ τώρα σε μερικά σημεία τα οποία ήθελα να τα τονίσω και θα ολοκληρώσω με αυτό. Οι προτάσεις μας για το μέλλον. Και που τις είχαμε υποβάλει εδώ και 1,5 χρόνο και που το Κοινοβούλιο ενέκρινε αφού τις μελέτησε αμελητή. Υπό την αιγίδα των προηγούμενων εισηγητών ήθελα εδώ να χαιρετήσω το έργο τους, το ρόλο τους και να πω ότι ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι τη δράση και να έρθει σε διάλογο με το Συμβούλιο όσο το δυνατόν συντομότερα. Το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω και να αναφέρω είναι η άοκνη προσπάθειά μας να ε, σχεδιάσουμε έτσι την πολιτική που να μπορέσει να διατηρηθεί σε όλη την επόμενη δεκαετία. Έχουμε εδώ μια στρατηγική επιλογή. Έχουμε προτείνει μια πολιτική που θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη για όλες τις περιφέρειες και τις περιοχές της Ευρώπης. Και πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ καλούς λόγους να είμαστε θετικοί για την πολιτική μας αυτό που ονομάσαμε δίδυμη μετάβαση. Twin transition. Θα πρέπει ως Ευρώπη να το ενστερνιστούμε, διότι είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον της Επίρου και για τη συνοχή μας στην Ευρώπη. Αυτή η διπλή, η δίδυμη λοιπόν, μετάβαση έχει να κάνει με την τεχνολογική επιτάχυνση και την κλιματική μετάβαση. Η ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη έχει αναγγείλει κάποια πολύ σαφή μέτρα. Κατά δεύτερον, και το λέω μόνο και μόνο για να το καλύψω, υπάρχει και αυτό το αναθεωρημένο μενού ευρύτερων, σφαιρικότερων πολιτικών στόχων. Κατά τρίτον, προτείνουμε να επικεντρώσουμε πολλά από όσα ήδη διαθέτουμε στις πρώτες μας προτεραιότητες για την Ένωση και από γενική σκοπιά και από την πλευρά της συνοχής της ίδιας. Προτείναμε να επικεντρωθούμε στο να διασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος στην Ευρώπη με την καλύτερη διασπορά της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και άρα η συνοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί και σε αυτούς τους πολιτικούς στόχους παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Κατά δεύτερον, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στους πολιτικούς στόχους διότι αυτό ταυτίζεται με τους στόχους μας της κλιματικής ε, αλλαγής. Σας ανέφερα την κυρία Φόντερ Λάιεν. Έχει πει, όπως γνωρίζετε, ότι θεωρεί ότι πρέπει τους στόχους μας για το 2030 να τους αυξήσουμε. 50% περικοπή των εκπομπών διοξιδίου του θερμοκηπίου, διοξιδίου του άνθρακα τουλάχιστον. Όμως 2030 είναι η επόμενη περίοδος προγραμματισμού. Εκεί πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Και νομίζουμε ότι στις μεσοποτάσεις που κάναμε να επικεντρωθούμε στην πολιτική συνοχή και σε αυτόν τον πολιτικό στόχο, κάτι ε, θα πετύχουμε. Μια βιωσιμότερη και πρασινότερη Ευρώπη. Και τέλος, ε, στα πλαίσια του εξυγχρονισμού αυτού, του φρεσκαρίσματος, να θυμίσω και πάλι την πρότασή μας για μια προσέγγιση 5 συν στον προγραμματισμό. Θεωρούμε 5 συν 2. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους η ευελιξία είναι απαραίτητη για να μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες της τελευταίας διετίας πάντοτε, ανάλογα με το ρού των γεγονότων και ανάλογα με την μετάφραση και το κατά πόσον θα έχει πετύχει. Σε ε, πέντε χρόνια από τώρα θα υπάρχει άλλο κοινοβούλιο, νέα θητεία, άλλη επιτροπή και προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε και τα απρόπτα. Όντως θέλουμε την απλούστευση. Χαρήκαμε πολύ που η προσπάθειά μας να πάμε όσο μακρύτερα γίνεται με την απλούστευση έχει αποδώσει καρπούς και την απεδέχθησαν οι συνομοθέτες. Βλέπουμε όμως να υψώνεται και ο φόβος που είχαμε και προηγουμένως. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τα πράγματα περιπλέκονται ξανά και εδώ να θυμίσω να μην λησμονήσουμε τον σημαντικό αυτό στόχο απλούστευσης που ήδη είχαμε αρχίσει να επιδιώκουμε και είναι σημαντικός. Τρίτον, η εκκλησία μου νομίζω έχει γίνει κατανοητή. Πρέπει να βιαστούμε δεν έχουμε αρκετά γοργά αποτελέσματα για τους πολίτες. Δεν μπορούν να μας περιμένουν. Η πολιτική συνοχή πρέπει να ε, λειτουργήσει, να βρεθεί εκεί που πρέπει για να επιτρέψει την ε, μετάλλαξη σε κάποιες περιπτώσεις, την ε, αλλαγή και να μπορέσουν οι πολίτες να γίνουν οι ίδιοι κύριοι αυτής της αλλαγής. Το παιχνίδι το έχουμε παίξει και στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τους ρυθμούς, να το κάνουμε και στο μέλλον. Όπως θα είδατε, ακούσαμε πολλά που μπορούν να επιτρέψουν την επιτάχυνση της πολιτικής δράσης. Δεν είναι μόνο ένα, δύο ή τρία πράγματα. Πρέπει να υιοθετήσουμε προγράμματα εγκαίρως. Όχι 12 ή 18 μήνες καθυστερημένα. Ε, έχει να κάνει με τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη σε αυτή την περίοδο να συνεχίσουν αμέσως χωρίς καθυστερήσεις στην επόμενη περίοδο. Να μην χάσουμε χρόνο αυτό το σταμάτα ξεκίνα που διαρκώς ε, δημιουργεί προβλήματα. Ούτε χρειάζεται να επινοήσουμε εδώ τον τροχό. Είναι προγράμματα που ήδη είναι σε εξέλιξη σήμερα να συνεχίσουν. Αυτό θέλουμε απλώς. Ο δρόμος έχει ανοίξει να τρέξουν. Και Τέλος, το τρίτο που θέλω να πω είναι ε, η δικαιοσύνη. δηλαδή να επικεντρωθούμε στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, οι προτάσεις μας στηρίζουν τις περιοχές αυτές, αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ της αλληλεγγύης για τις φτωχότερες περιοχές και της ανάληψης ευθύνης από τους ίδιους τους υπεύθυνους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν στην πράξη, λόγω χάρη στην συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να αναλυφθεί περισσότερη ε, ευθύνη από τα κράτη-μέλη για τα προγράμματα, από τους αρμοδίους σε εθνικό επίπεδο για την χρηματοδότηση και εκεί η πολιτική συνοχής θα έχει και περισσότερο πάτημα και μόχλευση και περισσότερη δυνατότητα επενδύσεων. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά ήταν ε, εξαντλητική και ειλικρινέστατη η παρουσίασή σας. Αλλά δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από σας. Θα δώσω το λόγο σε όσοι το ζήτησαν, με τη σειρά που τον ζήτησαν. Πρώτα η κυρία Κορίνα Κρέτσου, μετά η Κωνστάς Κρέλ και παρακαλώ τη γραμματεία να καταγράψει και τους υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτα οι συντονιστές, αλλά πριν τους συντονιστές η Κορίνα Κρέτσου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά Λεμέτ, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την ε, σκληρή δουλειά που κάνατε ε, στις υπηρεσίες σας, στην ε, Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Είχαμε εργόδεις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, πολύ σκληρό τιτάνιο έργο. Τώρα είμαι πια ευρωβουλευτής και έχω αλλάξει στρατόπεδο. Ο ρόλος μου θα είναι να είμαι σκληρή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά νομίζω ότι στόχος μας είναι η συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προασπίσουμε το κοινό μας έργο. Όπως είπατε, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της εφαρμογής. Είχαμε πάει σε πολλα κρατημέλη και μαζί μερικές φορές πρωτοστατώντας ε, σε νέα σχέδια και επισπεύδοντας την εφαρμογή των προγραμμάτων. Λυπάμαι που βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα και θα πρέπει να ρωτήσουμε και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, που δεν εκταμείευσαν τα κονδύλια και που στέρισαν από τους συμπολίτε τους την ευκαιρία μιας καλύτερης ζωής και καλύτερου βιωτικού επίπεδου. Για να σας δώσω και ένα παράδειγμα από την πατρίδα μου, που, τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα. Από ό,τι ξέρω είναι βραδύς ο ρυθμός εφαρμογής και δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο ή πρόγραμμα που δεν έχει, δεν έχει υποβάλει ακόμη η Ρωμανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Που σημαίνει ότι έχουν παγώσει τα κονδύλια, δεν θα, διατεθούν, θα διατεθούν. Υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα, αλλά είναι στις Βρυξέλλες και περιμένουν επιλέξιμα προγράμματα. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν την ευθύνη και των κρατών μελών και να τα καλέσουμε να την επομισθούν. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις ε, για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Γιατί ε, ήταν δύσκολο το έργο μας και όπως είπε και ο Πρόεδρος ο μαζί και ενώπιον μας βρίσκονται χαλεπή καιροί, θέλουμε ε, ένα ισορροπημένο σχέδιο, ένα ισορροπημένο προϋπολογισμό και για πρώτη φορά έχουμε ε, 370 δισεκατομμύρια τον πιο γενναίο προπολογισμό των τελευταίων περίοδων, θα πρέπει να δώσουμε μάχη γι' αυτό. Ε, μέχρι τις 2 ε, Μαΐου είχαμε μόνο τρεις τριμέρες διαλόγους και ήταν πραγματικά μυστήριο για μένα γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθυστερεί τόσο σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ και σε 1,5 χρόνο μόνο μία φορά ενέκυψε το ζήτημα αυτό που είναι τόσο σημαντικό του ΠΔΠ. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι τα περισσότερα κράτη, πάνω από 10 χώρες, ε, ε, περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζονται στα κονδύλια αυτά. Πάνω από το 50% των δημόσιων επενδύσεών τους ε, προέρχεται από αυτά τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Οπότε είναι και όφελο του Συμβουλίου να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσει για το πει. Θα πρέπει να συστήσουμε ένα κοινό μέτωπο, λοιπόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης. Και ευχαριστώ τους πρώην και νυν ευρωβουλευτές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και στην προηγούμενη θητεία. Και είμαι σε κάπως περίεργη θέση τώρα, ε, από Επίτροπος Ευρωβουλευτής. Πάντως, κύριε Λεμέτρε, μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς όφελος και προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κρέτσου. Ο κύριος Νοβάκοφ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Κύριε Λεμέτρ, αγαπητέ Μάρκ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα και εγώ να σε καλωσορίσω σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά τις θερινές διακοπές και χαίρομαι που ξεκινάμε με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Μας παρουσίασε ε, μια ομιλία που δείχνει πόσο που είπε ότι ε, δείχνει ότι είσαι και όχι πολιτικός, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Διαφωνώ όμως, γιατί έχεις ε, αίσθηση και γνώση του πόσο σημαντικός είναι ο κανονισμός αυτός για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική συνοχή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις λοιπόν γνώση και πολιτική γνώση του πράγματος εκτός από την τεχνική. Πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ για τις προσπάθειές σου και παρακολουθώ το έργο σου εδώ και πολλά χρόνια. Στην αρχή είχα αποφασίσει ότι η καμπύλη των επιδόσεων ήταν περίπου 100% και σκέφτηκα καλό αυτό. Μετά όμω ε, διαπίστωσα ότι είναι το μισό, το 50% ε, των επιδόσεων. Και μερικέ χώρε είναι στο μισό του μισού, δηλαδή στο 25% των ε, αναμενόμενων επιδόσεων. Και πραγματικά αυτό είναι ανησυχητικό, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Γιατί πέντε χρόνια μετά την έναρξη τη περίοδου προγραμματισμού είμαστε σε τόσο χαμηλό ποσοστό. Τα βλέπω κάπω σκούρα εδώ και μάλιστα τη στιγμή που εξετάζουμε το μέλλον του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και νομίζω ότι όλοι εμείς οι φίλοι της πολιτικής συνοχής θα ζητήσουμε περισσότερη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Και από τη στιγμή που αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί μόνο το 25% των κονδυλίων έχουμε εκταμιεύσει. Πώς θα διεκδικήσουμε λοιπόν αύξηση ενώ δεν έχουμε καταφέρει να εκταμιεύσουμε τα διαθέσιμα πολύ φοβάμαι ότι γνωρίζω την απάντηση αν διεκδικήσουμε πιο δαψίλη προπολογισμό. Έχω μια απλή και σύντομη ερώτηση. Είπες, ε, είπατε ότι είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις και εγώ ως ε, ε εισηγητής για το CPR και εγώ είμαι έτοιμος, αλλά το Συμβούλιο πιστεύετε ότι είναι έτοιμο. Γιατί εμείς εδώ και έξι μήνες είμαστε έτοιμοι. Το Συμβούλιο όμως κόλλησε η εργή και δεν κάνει ένα βήμα εμπρός. Ξέρω τι προσπάθειες έκανε η Επίτροπος Κρέτσου και η συνεισηγήτριά μου, η κυρία Κρέλ. Αν όμω πάμε προς την, αυτή, προς την κατεύθυνση αυτή, με την ίδια ταχύτητα, η περίοδος προγραμματισμού 21-27 δεν φαίνεται, δεν προδιαγράφεται καλύτερη από την τωρινή. Άρα έχω δύο ερωτήσεις. Πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι τους τριμέρους διαλόγους με πλήρη εντολή του Συμβουλίου και δεύτερον, ποια μέτρα έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τις επιδόσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα ποσοστά απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές, κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις και για την σημερινή αλλά και για τη μελλοντική προγραμματική περίοδο. Κύριε Λεμέτρη, λέτε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχει καλή ροή των κονδυλίων και ότι υπάρχουν ποσά τα οποία δεν ε, ρέουν. Μιλήσατε για την γραφειοκρατία και από πλευράς της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει κάτι στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες θετικές ιδέες που μπορεί να έχουν ε, θετικές επιπτώσεις. Πώς ε, αυτή η απλοποίηση, η απλούστευση των διαδικασιών θα βελτιώσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρώ ότι αυτό που είπατε ότι πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων εξάντε η ε, θέση των κριτηρίων για την αιρεσιμότητα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά διαπιστώνω ότι στις προτάσεις της Επιτροπής αυτό έχει πάψει να ισχύει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν μου λέτε τι θα γίνει με το θέμα του αποθεματικού όσον αφορά δηλαδή τις επιδόσεις, τα κριτήρια που αφορούν τις επιδόσεις. Αυτό το αποθεματικό ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εκτός εάν υπάρξουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να αποσυρθεί αυτή η καινούργια πρόταση, το σχέδιο πρότασης. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, χρησιμοποιείται διαφορετικά, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, το πόσο αυτό που βρίσκεται στο αποδοματικό. Για πείτε μου ακριβώς αυτή η μεταρρύθμιση, τι αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή, έτσι και αλλιώς θα χρησιμοποιήσετε κάποιες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ή περιμένετε πρώτα να περάσει η πρόταση της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, ξέρετε πολύ καλά τι έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητά το 30% των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής να διατίθενται στο μέλλον για θέματα που αφορούν το κλίμα. Όμως ξέρουμε ότι την ίδια ώρα ζητούμε και περισσότερη ευελιξία για τις διάφορες περιφέρειες. Αν αποφασίσουν οι συναρμόδιες αρχές για την ε, νομοθεσία να ληφθούν υπόψη και κάποια τεχνικά προβλήματα, πώς εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν νέες ενδείξεις όσον αφορά τις ε, πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ξέρω πολύ καλά ότι όποια και αν είναι η πρόταση της Επιτροπής, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχτούμε αυτές τις ε, νέες προτάσεις. Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου ξέρουμε και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί και χωρίς συμφωνία η προοπτική ενός Brexit χωρίς συμφωνία δυστυχώς γίνεται πραγματικότητα. Τι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν εν ώψη αυτού του Brexit χωρίς συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συντονιστή μας, τον κύριο Κνότεκ, χρειάστηκε να πάει σε μια υπήγουσα υπόθεση του. παντού στην προεκλογική εκστρατεία και στην νησορειονιό, στον Ειδικό Ωκεανό, ε, είχα πολλές καλές συζητήσεις με συμπολίτε μου και παντού άκουσα, άκουσα την βεβαιότητα ότι η Ευρώπη είναι μια ευκαιρία, μια τύχη για τα εδάφια. Αλλά παντού άκουσα και την συστηματική μορφή, την αδυσόπιτη, αμήλικτη μορφή, ότι η Ευρώπη είχε γίνει σήμερα συνώνυμο της περιπλοκότητας. Ενώ για μας θα πρέπει η Ευρώπη να είναι συνώνυμο της εγκύτητας, γιατί αυτό προσπίζουμε εδώ και αυτό απαιτούμε εδώ. Απαιτούμε η πολιτική συνοχής οπωσδήποτε να είναι μια πολιτική που θα εξυπηρετεί τα εδάφη, τις περιφέρειες, τους κατοίκους. Και σήμερα επανειλημμένως ακούσαμε στην Επιτροπή μας την απέτηση του εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατικής Δομής. Είναι κατεπίγουσα λοιπόν η ανάγκη της απλοποίησης. Ερωτώ γι' αυτό. Ποιες είναι οι μέθοδοι που θα ακολουθήσετε ώστε η πολιτική συνοχή να γίνει πολύ πιο γρήγορα, πιο χρήσιμη και πιο αποτελεσματική για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και για τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες που ζούσε υπερπόντια διαμερίσματα 10.000 χιλιόμετρα μακριά από τις Βρυξέλλες και του Στρασβούργου, γιατί σήμερα αγαπούν ακόμη την Ευρώπη. Αν όμως στο μέλλον δεν τους συμπαρασταθούμε στον αγώνα τους κατά της απομάκρυνσης, της ε, περιθωριοποίησης, της απομόνωσης, θα μας γυρίσουν την πλάτη στο μέλλον και τότε θα τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η δημοκρατία. Και με την ομάδα μας, το Renew Europe, ε, εκεί βλέπουμε το μείζον διακύβευμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Στεφάν. Η συνάδελφος Μπαχομέα. Ευχαριστώ. Είμαι νέα Ευρωβουλευτής από τον Ιούλιο και παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την παρουσίασή σας. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την πατρίδα μου, την Ισπανία, σε ό,τι φορά το ποσοστό εκτέλεσης. Είμαστε πολύ κακοί μαθητές σε ό,τι φορά το ποσοστό εκτέλεσης. Γιατί, γιατί είναι ουραγός επιδόσεις η Ισπανία, υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια συγκεκριμένη αιτία, γιατί πραγματικά με θορύβησε αυτή η κατάσταση. Μπορείτε να με ενημερώσετε ή σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτή η και η κατάσταση για την Ισπανία σε ό,τι αφορά το ποσοστό απορρόφηση. Επίσης, μιλήσατε για τα σχέδια συγχρηματοδότησης ε, που θα είναι το κατάλληλο μέσο για να επισφευστεί η εκτέλεση των προγραμμάτων και των σχεδίων. Ερωτώ, υπάρχει δυνατότητα για συμπράξει σε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διεκπαιρέωση τέτοιων σχεδίων και προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή Ρέγγι, αλλά είμαι συνεισηγητής ε, για το ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Ε, αγνώμως τον συνεισηγητή μου από τους συλληστές δεν τον έχουν ορίσει ακόμη. Θα ήθελα να συνδέσω τη δική σας παρουσίαση με την παρουσίαση της μελέτης που ακούσαμε προηγουμένως και που αφορούσε τις νέες προκλήσεις και τις συστάσεις για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και το τι θα πρέπει να γίνει. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά σήμερα αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ο βαθμός εφαρμογής. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό σημείο, γιατί αν υπάρχει λυπής εφαρμογή, χαμηλό συντελεστής εφαρμογής. Το ενίσυν 3 είναι μία εξήγηση. Άλλη εξήγηση αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση στα κράτη-μέλη. Ασταθής πολιτική κατάσταση, ασαφής νομοθεσία. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να το δηλώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εσείς δεν είστε πολιτικός. Εμείς όμως είμαστε και μπορούμε να το πούμε. Και όταν βλέπουμε ποιες χώρες είναι στη χειρότερη θέση, η ερώτηση που προκύπτει είναι τι συμβαίνει. Προς τι, αν το είναι τρία ε, ισχύει για όλους, γιατί μερικές χώρες είναι ταχύτερες και άλλες βραδιπορούν. Αυτή είναι μια πολιτική ερώτηση που θα πρέπει να μας προβληματίσει και για τη μελλοντική συζήτηση θέλουμε και άλλες πληροφορίες για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και δεν χρειάζεται να δακτυλοδεικνύουμε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και να κατηγορούμε, αλλά να μην ε, θα ρίχνουμε όλα στον ίσυν 3. Επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Νοβάκοφ. Εγώ είμαι ο εισηγητή ε, για το ΠΔΠ και σα διαβεβαιώ ότι αυτή θα είναι η πρώτη μα αντίδραση. Όταν λέμε ότι θέλουμε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προπολογισμού για τη συνοχή. Και η πρώτη αντίδραση θα είναι, μα τι, να το κάνετε το ίδιο επίπεδο, αν είναι τόσο χαμηλό ο βαθμό εφαρμογή. Προ τι η διαφύλαξη του προπολογισμού. Ήδη και στο παρελθόν είχαμε τέτοια συζήτηση και θέλουμε επιχειρήματα για να στηρίξουμε τι απαιτήσει μα. Επίση, ε, το νησιν 3 δεν έχει επιπτώσει στην εφαρμογή μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στο Συμβούλιο δεν βιάζονται οι Υπουργοί. Το Συμβούλιο δεν βιάζεται λόγω του νησίντρια, γιατί γνωρίζουν ότι χρόνο υπάρχει. Οπότε όταν εμεί μιλούμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν έχουμε την αίσθηση ότι όλοι κόπτονται να το ε, οριστικοποιήσουν. Οι χώρε δεν βιάζονται καθόλου. Λέμε τέλη 2020, Γερμανική Προεδρία. Α, θα δούμε. Κάτσε και καρτέρα. Το νησιν 3 όμως ακριβώς ε, προβλέπει ότι τα νέα κονδύλια θα είναι για, τις, για τα παλιά προγράμματα για τα πρώτα τρία χρόνια, 2020, 2021, 2021 και 2023. Οπότε το νησιν 3 έχει έμπρακτες συνέπειες και θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί γιατί μεγάλο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και κατά του νησιν 2 και γι' αυτό θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι χαμηλό ο ρυθμό εφαρμογή, πού οφείλεται, πώ έχει κατάσταση στα συγκεκριμένα κρατημέλη. Θα πρέπει όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε. Και την τελευταία ερώτηση, ίσω κάπω προκλητική. Γιατί όπω πάντα προσπαθώ να είμαι προκλητικό. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε ότι υπάρχουν δύο πιθανότητε να καθυστερήσουμε παντού. Η μία πιθανότητα είναι να μην είναι έτοιμο το Συμβούλιο. Ότι δεν θα καταλήξει ομοφωνία στο εγγύς μέλλον στους επόμενους μήνες. Αυτό θα είναι μία αιτία της αργοπορίας. Να μην είναι έτοιμο το Συμβούλιο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα όλα θα αναβληθούν μέχρι τα τέλη του 2020. Δεύτερος λόγος αργοπορίας θα είναι ότι εμεί θα μπλοκάρουμε το Peter πει. Λάβατε το και αυτό υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πει όχι αν η πρόταση του Συμβουλίου δεν μα ικανοποιεί, μπορούμε να πούμε όχι στο πι. Γιατί το νέο Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι το σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πει όχι στο πι. Οπότε, αν πει όχι, τότε όλα θα καθυστερήσουν. Η ερώτησή μου είναι, τι πιστεύετε θα συμβεί στη συνέχεια, γιατί βλέπετε ότι στο Κοινοβούλιο αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αν έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, το Plan B που λέμε. Εσείς έχετε Plan B, έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο ή πιστεύετε το Συμβούλιο έχει τέτοιο Plan B, αν δεν είναι έτοιμο τα πράγματα το 2020. Δεν θα ήθελα να σας πω εμείς τι πιστεύουμε, γιατί τώρα το εκπονούμε αυτό το Plan B, την εναλλακτική μας λύση, την θέση αναδίπλωσης, αλλά ρωτώ και εσάς, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τέτοιο Plan B. Ε, θα ήθελα όλοι όσοι κρατούν τα πρακτικά να σημειώσουν αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Γιάνν Ολμπράιτ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Σόκολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λεμέτρα, και εγώ σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι και εγώ νέο μέλος ανήκα στο Κοινοβούλιο της Κροατίας και έχω παρακολουθήσει κάποιες από τις συζητήσεις που αφορούν τα θέματα αυτά. Ιδιαίτερα όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στηριχθεί από το Ταμείο Συνοχής και αφορούν καινοτομία και έρευνα. Για λόγους τους οποίους αναφέρεται όπως θέματα που αφορούν μετανάστευση, μετατοπίσεις πληθυσμών, διασυνοριακές περιοχές. Στην ε, Κροατία όχι το 50% αλλά το 80% τέτοιων προγραμμάτων ε, χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή, από τα κονδύλια αυτά. Αυτό είναι φυσικό. Είμαστε το τελευταίο κράτος που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλω εδώ να υπογραμμίσω είναι ότι ο κύριος σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής συνοχής της είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να πλησιάσουν το μέσο όρο και τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές. Από την άλλη, αν κοιτάξουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις χρηματοδότησης, αυτό που προτείνεται εδώ να πάμε από το νη συν 3 όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων στο νη συν 2, εδώ δεν νομίζω ότι ο σκοπός θα επιτευχθεί. Αν κατάλαβα καλά, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και κράτη-μέλη έχουν και τα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την συγχρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο το νη να παραμείνει. Και εδώ αναφέρομαι στη χώρα μου, στην Κροατία, οι δυνατότητες που διαθέτουν οι δικές μας περιφέρειες, τα κράτη μας, και εγώ μιλώ σαν το πιο καινούριο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο περιορισμένες. Και δεν ξέρω αν τόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μας σίγουρα θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και τον ίσιν 3 νομίζω δεν πρέπει να αλλάξει. Η απλούστευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για συνέργειες. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές πρόοδοι. Το Horizon, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τους κανόνες που αφορούν τη βελτίωση του ανταγωνισμού. Και βεβαίως πολλές φορές η σύγκριση μεταξύ περιοχών και μεταξύ κρατών δείχνει τις τεράστιες διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε συγκεκριμένα βήματα, ενίσχυση της συνέργειας των συνεργασιών και για ποιο λόγο Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα υλοποίησης, χώρες που καθυστερούν. Ίσως χρειάζεται περισσότερη απλούστευση και πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα στα κράτη-μέλη τι συμβαίνει, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό. Είπατε ότι και αυτός ο τομέας έχει σημαντικές καθυστερήσεις σε κάποιες χώρες. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν συγκεκριμένα βήματα, να επιταχύνουμε τους ρυθμούς σε κάποια κράτη-μέλη και το νησιν 3 που θα γίνει νησιν 2 κάποια μέρα, τότε θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Μιλήσατε και για τη βιωσιμότητα, πάρα πολύ σημαντικός τομέας για όλες τις πτυχές ε, της ε, δραστηριότητάς μας και όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και άλλους τομείς που προσπαθούμε να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε συνέργειες και ευνοϊκά αποτελέσματα για τους πολίτες Μου Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λόπε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε το Γενικό Διευθυντή εδώ μαζί μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας παρουσίασε. Έχουμε εδώ εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας εξηγούν ότι όλα πάνε καλύτερα μεταξύ του 2014-2020. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εάν καταφέρουμε να φτάσουμε στο 50% απορρόφησης μέχρι το τέλος αυτής της προγραμματικής περίοδου, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά. Παρόλο που κάποιες χώρες δεν θα μπορέσουν να φτάσουν και να υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Όμως η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης είναι η πολιτική συνοχή. Αυτό το ξέρουμε στην Ευρώπη και η επιθυμία λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών να προχωρήσουν με καλύτερους ρυθμούς και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής συνοχής. Η απορρόφηση λοιπόν των κονδυλίων, η μείωση της τάξεως του 10% που θα είναι ο άμεσος αντίκτυπος του Brexit, είναι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και την Άνοιξη ψηφίσαμε δύο φορές για να παραμείνουν αμύωτα τα επίπεδα χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την τελική συζήτηση για το θέμα αυτό για ένα χρόνο. Δεν είμαστε λοιπόν καθόλου σίγουροι ότι η επόμενη συνάντηση κορυφής το Δεκέμβριο σύνοδος κορυφής, συγγνώμη, το Δεκέμβριο, θα πάρει μια σαφή απόφαση όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι οι επιθυμίες μας, αλλά πρέπει να περιμένουμε και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να διαμαρτυρόμαστε για το τι δεν πετύχαμε στο παρελθόν. Καλύτερα θα ήταν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον και είμαι πεπισμένος ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στείλουν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα παραδείγματος χάρη για αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό είναι, αν θέλετε, το καθοριστικό, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η δική τους ευθύνη και να αποφασίσουν αν ναι ή όχι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα ποσά αυτά αργότερα. Καλό θα ήταν τουλάχιστον το 2023-2024 να ξεκινήσει η χρήση αυτού του αποθεματικού και όλα τα κονδύλια να μπορούν να απορροφηθούν για το σκοπό για τον οποίο είχαν προγραμματιστεί. Το ερώτημα για μένα είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Μείωση της τάξης του 10%? Ο προϋπολογισμός θα μειωθεί στο 70% σε σχέση με το σημερινό προϋπολογισμό. Αυτό θα είναι πολύ κρίμα για τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα αποθαρρύνει τα κράτη-μέλη όσον αφορά το δικό τους κομμάτι της προσπάθειας. Ίσως θα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύστημα, ένα νέο μηχανισμό για να στηρίξουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες έτσι ώστε να φτάσουν σε καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερη ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους εάν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Το 2016 η περιφερειακή ανάπτυξη ουσιαστικά βασιζόταν σε μηχανισμούς και συστήματα τύπου ΝΑΤΣ. Η Λιθουανία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες σήμερα έχουν ενσωματωθεί σε μια άλλη κατηγορία. Αν κατάλαβα καλά, η πολιτική συνοχή είναι η καλύτερη, το καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για να μειώσουμε τις μεγάλες διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και να υπάρξει πραγματική εσωτερική και εξωτερική σύγκληση. Πιστεύω πραγματικά ότι όλη αυτή η αναταξινόμηση που έγινε το 2016 δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τις νέες προβλέψεις και προοπτικές ιδιαίτερα για την περίοδο ως το 2017. Εάν δεν κάνουμε ο καθένας αυτό που πρέπει για να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες, δεν θα μπορέσουν οι περιφέρειές μας να αναπτυχθούν. Κοιτάξτε την περιοχή Μαζορέσκη η οποία, εάν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, παραμένει σε επίπεδα φτώχειας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη δική μου χώρα, στη Λιθουανία. Η πρωτεύουσα, Βίλνιος, απορροφά το 11% ουσιαστικά των ε, κονδυλίων και μόνο 63% των κονδυλίων μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι οποίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα ή επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Αυτή λοιπόν η κατασταση τους αυτη λοιπον η αναταξινομηση που έγινε το 2016 νομίζω ότι δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τις μελλοντικές προοπτικές για τις οποίες θα πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Διευθυντή που είναι εδώ για να κινήσουμε και αυτή τη θητεία στο Κοινοβούλιο με καλή δουλειά, όπως και στην προηγούμενη θητεία, θέλω να το τονίσω και νομίζω ότι θα έχουμε τριμερείς διαλόγους για τρία σημαντικότατα ντοσχέ που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή. Η αντιπροσωπεία μου από το κίνημα των πέντε αστέρων έχει ήδη εκτιμήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά ακόμα περισσότερο μας ικανοποιεί που το κοινοβούλιο αυτό το περασμένο Μάρτιο είπε όχι ε, με καμία εξαίρεση στα ορυκτά καύσιμα. Οπότε θα έχουμε τώρα την ευθύνη να φέρουμε εις πέρα σε αυτήν την απόφαση. Και στην Ολομέλεια για το CPR, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται την ε, πρικοδότηση από τον προπολογισμό. Αυτό ζήτησε τουλάχιστον γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε περικόψει 2 ε, εκατομμύρια και εμείς ζητάμε να επιστρέψουμε στα 368. Είναι σημαντικό οι μεταφορές αυτές να γίνουν και από το, ε, από το 2020 και από το CLX. Και εδώ θέλω να κλείσω με μία ερώτηση και μία ευχή. Για την αιρεσιμότητα και την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Είναι σημαντικό για το Ευρωκοινοβούλιο αυτό και ελπίζω να έχετε υπόψη ποιε είναι οι διαπραγματευτικέ μα θέσει και να ενωθούμε, γνωρίζοντα τι ε, αντιρρήσει που είχαν προβάλει η Ισπανία και η Πορτογαλία στην περασμένη θητεία. Οπότε έτσι θα φτάσω στην ερώτησή μου. Στο ενοποιημένο κείμενο, δειλά το Κοινοβούλιο ζήτησε να ξαναδούμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Μαθαίνουμε τώρα από πηγές του τύπου ότι μπορεί να υπάρξει μια επαναθεώρηση κάποιων κριτηρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμφωνό Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μήπως πρέπει να δούμε τη διασπάθηση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων σε επίπεδο διευθυντικών ταμείων και πολιτικής συνοχής στα εθνικά κράτη και να δούμε πως αυτό ευθύνεται για τα ελλείμματα. Θα πρέπει να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση, λέτε. Πολύ ωραία, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο έλλειμμα, εφόσον τα κατημέλη στηρίζουν με τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Επίσης για τον κανόνα νη συν 3. Πολλές φορές λέμε ότι δεν γίνονται αρκετές δαπάνες από τα κράτη-μέλη. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια χαλαρότητα από πλευρά κάποιων συγκεκριμένων περιφερειών. Ωστόσο, δεν άκουσα να γίνεται λόγος, ε, ούτε να αναλαμβάνονται ευθύνες από τους ε, υπευθύνου όταν ορισμένες περιοχές και περιφέρειες δεν έχουν αρκετό δυναμικό στη διάθεσή τους, αρκετό κόσμο, δεν έχουν περιθώριο να κάνουν σωστά τα προγράμματά τους, ούτε ε, μπορούν οι τελικοί δικαιούχοι εύκολα να έχουν πρόσβαση στα ε, μέσα χρηματοδότησης. Ο ΦΠΑ είναι ένα κόστος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν λάβει ε, μέτρα και γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να προσέχει λίγο καλύτερα ε, για το πώ γίνονται οι δαπάνε τη τεχνική ε, στήριξη από τι περιφέρειε. Θα έλεγα να συγκεντρώσουμε καλύτερα πληροφορίε, όχι γενικώ και αορίστω για τα κράτη-μέλη αλλά ανακατηγορία περιφέρεια. Αν σκεφτώ τη χώρα μου, την Ιταλία, δεν μπορώ να πω ότι όλε οι περιφέρειες έχουν το ίδιο επίπεδο δαπανών, είναι βέβαια ότι οι νότιες περιοχές, οι περιοχές του Νότου, έχουν ε, χαμηλότερο επίπεδο εξόδων από τον Βορρά. Άρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνει σωστά μια διάκριση, μια κατηγοριοποίηση για να καταλάβουμε και καλύτερα πού πρέπει να πάμε να παρέμβουμε. Επίσης ακούστηκε ότι είναι άριστα τα αποτελέσματα γιατί υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, σχεδόν 430.000 νέες θέσεις. Τι είδου θέσει εργασία όμω είναι αυτέ. Ε, αορίστου, απεριορίστου διαρκείας, με βάουτσερ και δελτία, ε, part-time, τι δουλειέ λέμε και εννοούμε. Και ήθελα δύο ε, απαντήσεις. Λέτε για το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Το είπε και η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που Ήθελα να μου πείτε τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι project και πώς δεν θα πληγεί ε, που δεν είναι η πολιτική συνοχή από αυτή την ιδέα. Και επίσης, έχετε πληροφορίες, γιατί νομίζω ότι ήδη από τον Απρίλιο ακούγονται κάποια πράγματα, για την πιλωτική δράση της περασμένης Επιτροπής σε σχέση με τη βιομηχανική μετάβαση, όπου θα έπρεπε να συμμετέχουν 7 κρατημέλη και με τις περιφερειές τους. Η Επίτροπος Κρετού είχε ξεκινήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, μας το είχε παρουσιάσει. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο να έχουν προχωρήσει οι δράσει αυτέ, τι αποτελέσματα υπάρχουν και αν υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουν δημόσιε προμήθειε τη... με τη συμμετοχή νέων περιφερειών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ταμάντο. Και τελευταίο ομιλητή, η ομιλητρία μάλλον, κυρία Γκίζ. Μία ερώτηση για κάτι το οποίο ήδη έχει αναφερθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που για κάποιες περιοχές ε, με ορυχεία, ανθρακορυχεία δίνει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα σήμερα το γεγονός των ποσών που θα διατεθούν για την προστασία του κλίματος. Θα ήθελα να μου πει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν λαμβάνει υπόψη της τις δύο αυτές διαφορετικές κατευθύνσεις των χρηματοδοτήσεων στο νέο της προγραμματικό ε, προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα πάντως να σας πω κύριε Λεμέτου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Εμείς έχουμε ε, συγκεκριμένη πρόταση και είμαστε οργανωμένοι και μπορούμε να συνεχίσουμε τους τριμέρεις διαλόγους. Ήδη λάβαμε τα μέτρα μας ε, και έχουμε κλείσει και αίθουσες. Οπότε περιμένουμε σήμερα την αντίδραση του Συμβουλίου. Και μάλιστα ήρθατε μετά από μια ανταλλαγή απόψεων που είχατε με τη Φιλανδική Προεδρία και διαπιστώνω δυστυχώς ότι ε, ζητούμε από εσά απαντήσεις ενώ το Συμβούλιο έδωσε ελάχιστες απαντήσεις. Μέχρι στιγμής δυστυχώς το Συμβούλιο έχει δείξει ότι δεν επιθυμεί να οργανώσει άτυπο Συμβούλιο για την πολιτική συνοχή ε, όπως ήθεστε, από όλες Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άκουσα ότι ακόμη και το θέμα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων αμφισβητείται, αν θα γίνει. Οπότε διαπιστώνουμε σημαντικές δυσκολίες εκ μέρους του Συμβουλίου. Και δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα επανέλθει στους τριμέρις διαλόγους. Ήσασταν στο τελευταίο τριμέρι διάλογο και εκεί ε, καταγράψαμε κάποιες άτυπες συμφωνίες. Και πραγματικά ελπίζω από βάθος καρδίας ότι το Συμβούλιο ε, θα επανέλθει στους τριμερείς διαλόγους ε, με βάση τις ε, συμφωνίες που ήδη έχουμε καταγράψει. Και σας διαβεβαιώ ότι σήμερα είστε απέναντι σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει στεναρές αποφάσεις και θα προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με σταθερό και επικοδομητικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι το επίπεδο εφαρμογής δεν μας βοηθά στις διαπραγματεύσεις και δεν στηρίζει τα επιχειρήματά μας. Πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Όλμπριχτ ότι χρειαζόμαστε επιχειρήματα για να αντισταθούμε στις επικρίσεις που μας απευθύνονται. Βέβαια, ξεκινήσαμε τα προγράμματα με μεγάλη καθυστέρηση καταρχήν. Εν συνεχεία, περάσαμε σε άλλο σύστημα. Αλλάξαμε σύστημα με σημαντικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτό για τις περιφέρειες. Ούτε και αυτό μας βοήθησε στην σωστή αξιοποίηση των κονδύλων. Και θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες για τα κράτη-μέλη. Με αποτέλεσμα να έχουμε επιπλοκές σε επίπεδο περιφερειών για την απρόσκοπτη αξιοποίηση των κονδύλιων. Και αυτό το λέω για να αποποιηθούμε των ευθυνών μας ε, ή για να απαλλάξω κανέναν από τις ευθύνες τους. Αλλά αυτό είναι, αυτά είναι αντικειμενικά περιστατικά που δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό τις καθυστερήσεις. Φυσικά περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις και τα δικά σας σχόλια για να δούμε πώς μπορούμε να υπερβούμε τα προσκόμματα που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτή την περίοδο, να τα αποφύγουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης, μία ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το αναφέρατε κι εσείς. Όντως, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο παίζει σήμερα όλο και πιο σημαντικό ρόλο και ίσως το μέλλον να έχει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο και ενισχυμένο. Πώς λοιπόν η Γενική Διεύθυνσή σας, η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, εντάσσεται στη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, και πώς συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟΦΗΝ. Είστε σε θέση να υποστηρίξετε τις ε, περιφέρειες ε, όταν αυτό χρειαστεί και απέναντι στη Γενική Διεύθυνση Εκοφήν. Αυτά είναι 5,5. Έχετε χρόνο, έχετε κρατήσει και σημειώσεις και προλαβαίνετε να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας ε, για την πολύ πλούσια συλλογή σχολείων και ερωτήσεων που με επιτρέψετε να συγκεντρώσω. Και παρόλο που έγιναν πολλά κοινά σχόλια, θα προσπαθήσω με συστηματικό τρόπο να διατρέξω τις παρατηρήσεις σας και να καλύψω το σύνολο των θεμάτων που θίξατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το σχόλιο της κυρίας Κρέτσου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ισχύει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ε, έχει αναδείξει το ΠΔΕΛΤΑΠΗ ως βασική του προτεραιότητα. Πάντως ευελπιστούμε ότι από τον Οκτώβριο και μετά όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει μια πιο ευρυθή συζήτηση για το ΠΔΠ. Ευελπιστούμε ότι τότε θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένα σχόλια και θα περάσουμε σε μια πιο αποφασιστική φάση. Και εσείς και εμείς ε, διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής το έργο του Συμβουλίου περιστράφηκε σε πολύ γενικά ζητήματα. Τίποτα συγκεκριμένο, συγκεκριμένη αριθμή. Έχουμε βέβαια την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σε αντίθεση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι σαφή και ποσοτικοποιημένη, στο Συμβούλιο δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο νούμερο. Δεν υπάρχει καν ψαλίδα, φάσμα ποσών αριθμών. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει στο μέλλον στις επόμενες εβδομάδε ελπίζουμε η Προεδρία του Συμβουλίου να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιο ουσιαστική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, που ελπίζω να μην μονοποληθεί από ένα άλλο θέμα. Και ελπίζω να προλιάνει το έδαφος η Προεδρία του Συμβουλίου για την πιο ευρυθή συζήτηση, υποβάλλοντας ενδεχομένω και κάποιες προτάσεις, κάποιες ψαλίδες τουλάχιστον κονδυλίων ώστε να έχει κάτι πιο απτό, κάτι πιο συγκεκριμένο το Συμβούλιο για να συζητήσει. Και όχι μόνο γενικά και όριστα θέματα. Και εμείς εξακολουθούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετωπίζει σοβαρά τα συμπεράσματά του, ότι θέλει δηλαδή να υλοποιήσει τη συμφωνία για το ΠΙΔΕΛΤΑ μέχρι τα τέλη του έτους, γιατί αυτό αναφέρουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και ελπίζουμε να ισχύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπενθυμίσει στο Συμβούλιο αυτό το στόχο. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί μια ενδεχόμενη συμβαστική λύση, προτιμώ να μην κάνω προβλέψεις σήμερα, κυρία Κρέλ. Αλλά σίγουρα μπορείτε να υπολογίσετε σε εμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει στεναρά τις θέσεις της και τις προτάσεις της. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 χωρών, που θα είναι οικονομικά πιο αποδυναμωμένη μεν, θα χρειαστούμε νέους μηχανισμούς, νέα μέσα, περισσότερα κονδύλια σε κάποιους τομείς που δεν θα κατανομάσω τώρα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να συνεργαστούν και να συγκεντρώσουν κονδύλια, να τα μοιραστούν, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τα εφόδια να αντιμετωπίσουμε το μέλλον όπως θα έπρεπε. Και ε, για αυτό το σημείο χαίρομαι που με αντιληφθήκατε όταν εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για την παρούσα κατάσταση εφαρμογής. Καταρχήν, κάνω μια προσπάθεια υπέρ της συνοχής, που δεν προχωρεί όπως θα έπρεπε, όπως θα όφιλε. Αν είχαμε καλύτερη και ταχύτερη χρήση των διαθέσιμων ποσών, θα είχαμε μια πιο αποτελεσματική συνοχή. Και το πρώτο μας μέλημα είναι οι πολίτες, από τους οποίους ε, ζητούμε υπομονή. Αλλά στη συνέχεια έχουμε και την προάσπιση της ε, εικόνας της πολιτικής συνοχής, του κύρους της πολιτικής συνοχής. Και εκεί δεν είναι και πολύ ρόδινα τα πράγματα σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε 7 χρόνια από τώρα να είμαστε στην ίδια κακή κατάσταση, στην ίδια δύναμη θέση. Και ελπίζω ότι μετά από 7 χρόνια κάνουμε τέτοια συζήτηση, να είστε βέβαιοι ότι αν έχουμε παραμείνει σε κακή εφαρμογή, δεν θα έχουμε μόνο φίλου τη συνοχή Και αυτό είναι στρατηγικό ζήτημα και αφορά τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξέλιξη της πολιτικής συνοχής. Και θα ήθελα να σας πω ομά και ξεκάθαρα τι πιστεύω ακράδαντα. Αν δεν αλλάξουμε τον κανόνα νήσιν διάρκειας. Σας υπενθυμίσω, δεν προτιμούμε, δεν προτείνουμε βίαιη επαναφορά του νησί 2, αλλά σταδιακή και ομαλή. Αν δεν αλλάξουμε όμως το νησί 3, ό,τι απλούστευση και αν προτείνουμε, που προτείναμε, όσο και αν εξασφαλίσουμε συνέχιση του συστήματος και ούτω καθεξής, σας στοιχηματίζω ότι θα εξακολουθήσει να μείνει η εφαρμογή σε χαμηλά επίπεδα. Οπότε η αλλαγή του κανόνα νησι 3 είναι έτοιμα της λύσης. Αν θέλετε να συνεχίσετε σε βραδύ εφαρμογή, τότε κρατήστε το κανόνα νησι και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει τέτοια αργή εφαρμογή και στο μέλλον, ό,τι άλλες αλλαγές και αν κάνουμε στο σύστημα. Τώρα, και να ολοκληρώσω αυτό το θέμα, το θέμα του νησιν 3, του κανόνα νησιν Δεν άκουσα ποτέ κανέναν να μου εξηγεί με πιστικό τρόπο γιατί καταφέραμε να κλείσουμε τις δύο προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού με νησιν 2 και ξαφνικά τώρα δεν μπορούμε. Και το 2006 το κλείσαμε με το νησιν 2 και το 2013 το κλείσαμε με το νησιν 2 και τότε είχαμε περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα και τα κράτη-μέλη είχαν λιγότερη πείρα με την πολιτική συνοχή. Είχαμε 12 τότε νέες χώρες μέλη που έπρεπε να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχή και τα κατάφεραν με περισσότερα κονδύλια από ό,τι προτείνουμε τώρα και με τον ΙΣΙΝΔΙΟ. 2. Οπότε θα πρέπει να ψαχτούμε λίγο και τα κράτη-μέλη κυρίως για τον κανόνα αυτό. Και ξέρετε ότι πιστεύω ότι βάλουμε πολλά μέτρα που θα διευκολύνουν την ταχύτερη εφαρμογή στο μέλλον και θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την επίσπευση, την επιτάχυνση. Και δεν θα χάσουμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει μείωση των κονδύλιων στο μέλλον. Σε καμία περίπτωση. Θέλει απλώς αποτελεσματική πολιτική της συνοχής. Μια πολιτική συνοχής που θα υλοποιεί τους στόχους της προς το συμφέρον των συμπολιτών μας. Τώρα το Συμβούλιο είναι έτοιμο. Λυπάμαι που το ακούω απογοητευθήκατε από αυτά που είπε η... Ακούστε για την Προεδρία του Συμβουλίου. Και ήδη πριν το καλοκαίρι είχαμε άτυπες επαφές με την Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά και μαζί σας και με τη γραμματεία της Επιτροπής σας, ώστε το συντομότερο δυνατό, στις αρχές Σεπτεμβρίου δυνατόν, να συμφωνήσουμε για ένα πυκνό και φιλόδοξο πρόγραμμα συνεδριάσεων, άτυπων συνεδριάσεων, τυπικών συνεδριάσεων, τριμερούς διαλόγου, ώστε να καταλήξουμε σε όσο περισσότερα πιο κοινά σημεία γινόταν μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτός είναι κοινός μας στόχος. Και με βάση τις διμερείς επαφές που είχα και με την Προεδρία του Συμβουλίου, πιστεύω ότι και το Συμβούλιο συμμερίζεται αυτό το στόχο. Να καταλήξουμε έστω σε μερική συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Και θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο φιλόδοξο το Συμβούλιο, όχι μόνο να επιδιώκει μερική συμφωνία, αλλά ευρύτερη συμφωνία, συνολική, μακάρι. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα μέχρι το τέλος του έτους να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για όλα τα στοιχεία που είναι θεμελιώδη για τον προγραμματισμό και που είναι απαραίτητα για τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να χαράξουν το πρόγραμμά τους και να μας υποβάλουν προγράμματα που θα είναι συμβατά με το πιθανό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν έχω καμία ψευδέστηση για το κανονισμό περί κοινών διατάξεων, με το κανονισμό για το ενισχυμένο κοινωνικό ταμείο και το καθεξής δεν θα εφαρμοστούν πριν τα μέσα του επόμενου έτους, το νωρίτερο και κατά πάσα πιθανότητα προς τα τέλη του 2020 το βλέπω. Αυτό είναι τραγικό. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κανένα, κανένα δράμα, αλλά θα πρέπει το προγραμματικό τουλάχιστον σκέλος να το έχουμε έτοιμο νωρίς, νωρίτερα, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν πιο άνετε επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε μέχρι τα τέλη του έτου να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τα λειτουργικά προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα και να κερδίσουμε πολλά σε σχέση με την παρούσα περίοδο. Γιατί η χαμηλή εφαρμογή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως μας είπατε, στις πολλές αλλαγές που έγιναν στους κανόνες για την τρέχουσα περίοδο. Άλλαξε το σύστημα και στα κράτη-μέλη. Άρδιν. Χρειάστηκε μερικές φορές να ξεκινήσει εκ του το νέο σύστημα. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε καλή προετοιμασία έγκαιρη των προγραμμάτων. Με αποτέλεσμα τα προγράμματα να εγκρίνονται στα τέλη του 2014 ή μερικές φορές στα τέλη του 2015. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε αυτή τη φορά. Και πιστεύω ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αν βέβαια υλοποιήσουμε το στόχο το να ρυθμίσουμε όλα τα στοιχεία προγραμματισμού από το κανόνα περί κοινών διατάξεων και το κανονισμό για το Περιφερειακό Ταμείο μέχρι τα τέλη του έτους. Και ελπίζω στο εγγύς μέλλον να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ως προς το χρονοδιάγραμμα για τους τριμερείς διαλόγους, για τους επόμενους τριμερείς διαλόγους και να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, αν γίνεται. Κύριε Κρέλ, με ρωτήσατε για τα αποτελέσματα της επιπτώσης του κανονισμού Omnibus και τις προσπάθειες για την απλούστευση. Το επιδιώξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και μάλιστα μια πολύ πρόσφατη απόδειξη που προέκυψε πριν από λίγες μέρες και δεν είχε ακόμη υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, τώρα γίνεται αυτό, για πιθανή υποβολή ενστάσεων, γιατί πρόκειται για, τα, για πράξη, είναι να περάσουμε σε ένα καταποκοπή ποσό για την τεχνική αρρωγή. Ουσιαστικά προκαταλαμβάνει κάτι που είχαμε προτείνει για την μελλοντική περίοδο και επιτρέπουμε ε, σε προγράμματα να λάβουν χρηματοδότηση για ένα επιπλέον 4% για τεχνική συνδρομή. Κατά αποκοπή ποσό, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν τιμολόγια και ούτω καθεξής. Και αυτό προσπαθούμε να προτείνουμε στα κράτη-μέλη και ελπίζω να το δεχτούν. Πάντως μέχρι στιγμής δεν είδαμε και μεγάλο ενθουσιασμό να πετάνε τη σκούφια τους στα κράτη-μέλη για νέα πρόταση απλουστευμένο κόστος που προτείνουμε στον κανονισμό Omnibus. Με μία εξαίρεση. Και μάλιστα θα ήθελα να συγχαρώ το κράτος μέλος για αυτή την εξαίρεση, την Αυστρία. Η Αυστρία πραγματικά έδωσε το καλό παράδειγμα και προσπαθούμε σε συνεργασία με την Αυστρία να θεσπίσουμε ένα σύστημα ενεργειακής απόδοσης που επίσης ε, θα χρηματοδοτείται με βάση τον κανόνα ενός προκαθορισμένου ποσού κατά ποσού. Και αυτό θα το καταφέρουμε χάρη στο αρχικό όμνιμπους, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αυτό όμως θα πρέπει ε, να θεωρηθεί ως σπορά απλώς. Σπέρνουμε τώρα και θα δρέψουμε τους καρπούς την επόμενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό των επιδόσεων και την πρόταση που κάναμε εδώ και πολύ καιρό ώστε να μπορέσουμε να επαναπροσανατολίσουμε το αποθεματικό επιδόσεων για να χρηματοδοτήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Σας παρουσίασα την σχολαστική ανάλυση που κάναμε των επιδόσεων και στις συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη ακολουθούμε αυστηρά τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, το CPR, και ανακατανέμουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής το αποθεματικό των επιδόσεων. Βάση των προτάσεων των κρατών-μελών. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε επίπεδο υπουργών, ούτε τι απόφαση θα λάβει ή δεν θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποσυρθεί αυτή η πρόταση. που σε κάθε περίπτωση θεωρείται μη σκόπιμη. Για την επικέντρωσή μας σε συγκεκριμένα θέματα. Να πω σαφώς ότι δεν κλείνουμε τα αυτιά μας σε ιδέες όπως αυτές που ακούγονται στο Ευρωκοινοβούλιο που έχει φτάσει ως απόϊχος και στο Συμβούλιο ότι το να έχουμε περιφερειακή προσέγγιση και θεματική επικέντρωση είναι κάτι καλό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι εδώ δεν θα αποδυναμωθούν, δεν θα μειωθούν τα ποσοστά. Και τα τελικά ποσά που πηγαίνουν στην ευφιέστερη Ευρώπη και την βιωσιμότερη Ευρώπη. Και η Ευρώπη σίγουρα έχει πάρει αυτή την άγουσα. Για αυτούς τους δύο στόχους πολιτικής και ιδίως για τη θεματική επικέντρωση. Να επαναλάβω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι και πάλι να τονίσω τις δεσμεύσεις της Προέδρου της Επιτροπής για τους στόχους 2030 όχι να πάμε στο 40% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 90%, αλλά να φτάσουμε τουλάχιστον το 50% στο 2030. Κατ' εμέ, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί στον πολιτικό στόχο 2 να πάει κάτω από το ποσοστό της θεματικής επικέντρωσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσουμε εδώ τις φιλοδοξίες μας. Κάτι που το είχατε προτείνει μάλιστα εσείς οι ίδιοι ήταν ένας από αυτούς. Οι βιώσιμες αστικές μεταφοράς να περάσουν κάτω από τον πολιτικό στόχο 2. Αυτό χαμηλώνει τις φιλοδοξίες. Διότι ναι, Θέλουμε και βιώσιμε αστικέ μεταφορέ. Και ναι, αυτό θα, θα βοηθήσει την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ελπίζαμε όμω και ακόμη ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχημένη κλιματική δράση και βάσει άλλων πολιτικών στόχων. Και συγκεκριμένα δες μέσω των στόχων για τις μεταφορές, των πολιτικού, πολιτικού στόχου 3. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις με αμύωτο ενδιαφέρον και μάλιστα με κάποια ανησυχία. Πρέπει συνολικά να λάβουμε υπόψη τη νέα πολιτική ατζέντα της νέας επιτροπής, επί της οποίας το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει την κυρία Φοντερ Brexit. Πρέπει εδώ να διακρίνουμε μεταξύ του μέλλοντος και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για το άμεσο μέλλον, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, προετοιμαστεί διεξοδικός κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει και αποχώρηση, hard Brexit, χωρίς την παραμικρή συμφωνία. Η Επιτροπή θα σκύψει επί του θέματος αύριο ξανά. Δεν μπορώ να προδικάσω ότι θα αποφασίσουν αύριο Επιτροπή. Αλλά η Επιτροπή θα κοιτάξει για μια τελευταία φορά τα ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να προφυλαχθούμε κάπως, να βρούμε κάποια μαξιλαράκια και να αποκρούσουμε μερικά από αυτά που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Όλα δεν γίνεται να τα προλάβουμε. Να περιμένουμε λοιπόν αύριο την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής και να δούμε τι επιπλέον μπορεί να προτείνει η Επιτροπή αύριο. Θα επηρεάσουν και το τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και να πω και κάτι άλλο από την πλευρά της Επιτροπής ως μέρος των προετοιμασιών της. Θα είμαστε πανέτοιμοι να σκεφτούμε αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών εφόσον χρειαστούν, ιδίω για αυτά που θα πληγούν περισσότερο, και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να επανακατανείμουμε κάποιους πόρους βάσει των όσων τώρα ισχύουν στα τωρινά προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Και εδώ θέλω να πω στον κύριο Όλμπριχτ για το Plan B, το εναλλακτικό σενάριο. Νομίζω κανείς από εμά δεν θέλει να δει ως μια σοβαρή προοπτική, να ορθώνεται μπροστά μας το hard Brexit για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω εικασίες για σοβαρές καθυστερήσεις στην εξέβρεση συμφωνίας. Και εννοώ συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το ερχόμενο Πουδουπού. Έχουμε όλοι πολύ υψηλές και σοβαρές ευθύνες. Και με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο να λάβει θέση ως το τέλος της χρονιάς. Και μετά να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να καταλήξουν όλα τα θεσμικά όργανα σε μια συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι ουσιώδη σημασία για την Ένωση και είναι και σαφές ότι αν τα πράγματα στραβώσουν με το Brexit και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ε, χρησιμοποιήσει την πρόταση που δώσαμε εμείς προς το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να συμμετέχει και να συνεχίσει να συμβάλλει ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ακόμα και χωρίς ε, συμφωνία. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο στρέψει τα νότα του σε εμά, κατευθείαν σε εμά και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ταυτόχρονα, προφανώς θα έχουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρεώσεις και θα συνεχίσει να έχει υποχρεώσεις ακόμα και αν ξεκινήσει γυρνώντας την πλάτη σε μας. Πάντως, για τους ερχόμενους μήνες δεν θα ήταν επικοδομητικό να έχουμε συμφωνία για το Πουδουπού σε επίπεδο 27. Πάντως δεν θέλω να σκέφτομαι το Plan B. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Πρέπει η Ένωση να είναι πανέτοιμη και μάλιστα εγκαίρος. Να είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι με τα διάφορα κράτη-μέλη μας. Κύριε Μπιζού, Θα χρησιμοποιήσω τη φράση σας και ελπίζω να μην σας πειράζει. Περάσαμε όντω από την πολυπλοκότητα στην εγκύτητα, όπως το είπατε, ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι οι προτάσεις μας πηγαίνουν ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια κατηγορία προτάσεων που δεν τις ε, τόνισα. Ο πολιτικός στόχος 5 με τις ε, πλήρης της ε, ενιαίας δράσης σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο που η προσέγγιση εταιρική σχέση είναι όλος ιδιαίτερος ε, προαπαιτούμενη. Και εδώ το όριό μας ε, είναι ανύπαρκτο, είναι ο ουρανός όπως λέγεται. Το άπειρο εδώ για την ε, μελέτη που ανατέθηκε και την συμμετοχική προσέγγιση των πολιτών. Ο πολιτικός στόχος 5 αυτό ακριβώς επιτρέπει. Δεν πάμε να πούμε μέχρι πού πρέπει να φτάνει η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, στην επιλογή μεμονωμένων προγραμμάτων και project, αλλά οπωσδήποτε Η επιλογή διατίθεται στα κράτη-μέλη, προσφέρεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη, συμμετοχική προσέγγιση. Αν θέλουν, ας πούμε, να ανανεώσουν ή να φρεσκάρουν μια συνοικία, ένα πράστιο. Αυτός ο πολιτικός στόχος προσφέρει το ιδανικό πολιτικό πλαίσιο, το κατάλληλο πλαίσιο και την απαραίτητη ε, διαλλακτικότητα και ευελιξία, ώστε οι κάτοικοι μια ε, συγκεκριμένη συνοικία, ενό πλαστείου, να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, για αυτόν τον σκοπό. Όπω ξέρετε, προτείναμε να αυξηθεί το ελάχιστο επίπεδο συνεισφορά, μάλλον δαπανών, για αυτή την τοπική προσέγγιση από 5-6%. Εσεί προτείνατε να πάμε ακόμα παραπάνω. Δεν θα μα πείραζε και πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια προσέγγιση που πρέπει να ε, ε, εδρεωθεί και στην τοπική πραγματικότητα με μεγάλες φιλοδοξίες. Όσον αφορά τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και πέραν από την πολιτική συνοχής, θα αναφερθώ απλώς τις ανακοινώσεις που έχουμε ήδη κάνει και τις οποίες γνωρίζετε. Εμείς σαν υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμόδη για την οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση που καταφέραμε να επιβάλλουμε θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των διαφόρων εργαλείων, τα δημοσιονομικά εργαλεία και άλλα και φυσικά περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Κύριε Όλμπρεκτ. Μιλήσατε για την χαμηλή υλοποίηση, για τον ΙΣΙΝ 3. Νομίζω ότι αρκετά είπα για το θέμα αυτό. Θα συμφωνήσω με το επιχείρημά σας ότι πέρα από τις αρνητικές συνέπειες και την αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συζητήσει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αποδυναμώνεται γενικότερα η θέση μας εάν συνεχίσουμε με αυτά τα επιχειρήματα στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Σόκο, μιλήσατε για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, την χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων, εγώ βασίζομαι στην παρελθούσα εμπειρία μας. Γιατί σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και δεν έχουμε θέσει αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Το 2007-2013 ολοκληρώθηκε με τον συν 2 και με υψηλότερη κατανομή από αυτή που έχουμε σήμερα με νέα κρατημέλη που έπρεπε να εξοικειωθούν με το σύστημα. Και τελικά είδαμε ότι δεν υπήρχε σημαντική αποδέσμευση στο τέλος της χρονικής αυτής περίοδου. Και όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, μην ξεχνάμε την προϊστορία αυτού του τομέα. 87% αν θέλετε ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπήρχε πριν την κρίση, πριν το 2008-2009 με μεγάλη δυσκολία αλλά με επιτυχία πιστεύω βγαίνουμε από αυτήν την δεκαετή οικονομική κρίση και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι πλέον σημαντικό να επανέλθουμε στην ομαλότητα όσον αφορά την συγχρηματοδότηση και μια πιο ισορροπημένη κατάσταση μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. Το πιο υψηλό ποσοστό συγχρηματοδότησης ήταν 75%, όχι 85%. Όσον αφορά συνέργειες με άλλα προγράμματα, ναι, έχουμε σημειώσει την πολύ αυστηρή και επικριτική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνατότητες μεταφορών ποσών οι οποίες είναι ουσιαστικά μονόδρομος, δηλαδή βλέπουμε ποσά να βγαίνουν από την πολιτική συνοχή. Και τα μέτρα που προτείναμε έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική και να λειτουργήσει η δυνατότητα χρηματοδότησης με έναν ομαλό και απλό τρόπο, εύκολο τρόπο, κάποιες δραστηριότητες που τις ονομάζουμε προγράμματα αριστείας, δηλαδή κάποια προγράμματα και σχέδια πρωτοβουλίες που έχουν επιλεγεί βάση του Horizon και οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν ή να χρηματοδοτηθούν όταν δεν υπάρχουν εμπόδια κρατικής στήριξης από την πολιτική συνοχής. Κύριε Ρόπε, για τη μεταρρύθμιση του 2016 έχουμε επανέλθει στο θέμα αυτό και το συζητήσαμε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε νέα στατιστικά στοιχεία σήμερα. Πολύ καινούρια στοιχεία όταν έγινε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε στοιχεία για την ανεργία των νέων και έχουμε δύο νέα έτη για τα οποία γνωρίζουμε τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία και αυτό περιγράφεται σε ένα δελτίο που περιγράφει ακριβώς αυτές τις νέες πληροφορίες που διαθέτουμε και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Αυτή τη νέα πολιτική πρόταση η πολιτική συνοχή και τα ποσά πάντα λαμβάνουν υπόψη τα τελευταία, τα πιο επίκαιρα στατιστικά στοιχεία. Αυτή τη φορά, επειδή έχουμε πολύ πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και επειδή άλλαξε η κατάσταση, χάρη στην βελτίωση των τελευταίων ετών και την έξοδο από την κρίση, Γι' αυτό ακριβώς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό επιχείρημα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα τελευταία, τελευταία στατιστικά στοιχεία και να μην βασιστούμε σε μια θεωρητική πρόβλεψη. Ακριβώς γι' αυτό προτείναμε να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση των ΝΑΤΣ, όπως ακριβώς αναφερθήκατε, που σημαίνει μια αλλαγή για τη Λιθουανία, διάκριση της περιοχής του Βίλνιους, της πόλης του Βίλνιους από την υπόλοιπη χώρα και συγκεκριμένη προσέγγιση για την περιοχή του Μαζοβιένσκι. Ναι, όντως, αυτό είναι κάτι που προτείνουμε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο επ' αυτού. Πολύ συγκεκριμένα αναφέρθηκα στις εκθέσεις που αφορούν τις ε, χώρες μέλη. Έχουμε υπογραμμίσει στην έκθεση που αφορά τη Λιθουανία τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ε, περιφερειών της χώρας αυτής. Και υπάρχουν πολύ ανησυχητικές ε, διακυμάνσεις και διαφορές. 110% του μέσου όρου και κάποιες άλλες περιοχές που είναι στο ΝΑΤΣ 3. Με σοβαρά προβλήματα. Και ελπίζουμε οι αρχές της Λιθουανίας θα λάβουν υπόψη τους αυτά τα στοιχεία, γιατί σήμερα η Λιθουανία έχει ένα πρόγραμμα για όλη τη χώρα και δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ της περιοχής του Βίλνιους και της υπόλοιπης χώρας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια πιο λεπτομερής και εντελεχής εξέταση των στοιχείων που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των περιφερειών της Λιθουανίας. Κυρία Νταμάτο. Ψάχνω τις ερωτήσεις. Σύμφωνα σταθερότητα και ανάπτυξη. Ναι. Φαντάζομαι διαβάσατε πολύ πολύ προσεκτικά τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της α, κυρίας Βάντερ Λάιεν. Εξάλλου ήρθε και σας απίφθινε μια ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μίλησε για την χρήση εξ ολοκλήρου της ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης και σταθερότητας. Εγώ δεν είμαι από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ, που σίγουρα επεξεργάζεται όλες αυτές τις προτάσεις. Αυτό που είναι σαφές σήμερα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ανησυχητική κατάσταση. Βλέπουμε μια ύφεση οικονομική, μια επιβράδυνση των ρυθμών των οικονομικών και βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη μια χαλαρή νομισματική πολιτική. Υπάρχει ακόμα περιθώριο κινητοποίησης από μέρους της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίως φαίνεται ότι προετοιμάζει νέα μέτρα αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα επί της ε, οικονομίας. Τι άλλο μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και άλλα οικονομικά εργαλεία όπως η δημοσιονομική πολιτική και πώς μπορούμε να φτάσουμε στο κατ κατάλληλο οικονομικό μείγμα μέτρων, να ακολουθήσουμε δηλαδή και να συνοδεύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται από μέρους της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία αυτού του θέματος. Σημειώσαμε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις να ληφθεί υπόψη με έναν ιδιαίτερο τρόπο το θέμα της συγχρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο προγραμμάτων συνοχής. Το θέμα όμως ξεπερνάει αυτό. Πρόκειται για τις δυνατότητες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να δούμε τι άλλες δυνατότητες ευελιξίας υπάρχουν και να τις χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα. Όσον αφορά τα επίπεδα υλοποίησης, μιλήσατε για δυνατότητες περιορισμένες διοικητικής μεταρρύθμισης. Όντως υπάρχουν σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, σε κάποια τμήματα της Ευρώπης τέτοιες αδυναμίες και με τις Ιταλικές αρχές ξεκινήσαμε μια εταιρική σχέση για την ενίσχυση σε κάποιες Ιταλικές περιφέρειες των δυνατοτήτων της διοίκησης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, μακροχρόνια προσπάθεια. Αυτό δεν ρυθμίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται επιμονή για να βελτιωθεί η διοίκηση. Μιλήσατε όμως και για το παρελθόν, το 2007-2013, συγγνώμη, όπου οι Ιταλικές περιφέρειες ολοκλήρωσαν τελικά τα προγράμματά τους. Μιλήσατε και για το Μεσοτζόρνο, τον νότο της Ιταλίας. Και θα αναφερθώ σε μια ανησυχία που έχουμε και αφορά το θέμα της προσθετικότητας της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες και να κάνει τη διαφορά. Η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική παρά μόνο αν δεν υπάρχουν ταυτόχρονες περικοπές σε εθνικό επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων, της δημόσιας χρηματοδότησης. Και η τάση στο νότο της Ιταλίας είναι οι δημόσιες επενδύσεις σε μεγάλο βαθμό να μειώνονται και βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν. 0,4% του ΕΕΠ είναι στο νότο της Ιταλίας οι δημόσιες επενδύσεις και το επίπεδο αυτό δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να βοηθήσει την ανάπτυξη του, της Νότιας Ιταλίας και την σύγκληση της περιοχής αυτής. Αν συγκρίνει κανείς την αντίστοιχη επένδυση σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, φτάνουμε το 4%. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δεν... Εγγυάται λοιπόν αυτό το ποσοστό δημόσιων επενδύσεων καμία, με καμία έννοια την ε, προστιθέμενη αξία. Πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να κοιτάξετε με τις Ιταλικές αρχές αυτό το θέμα έτσι ώστε να βελτιωθεί τουλάχιστον στην τελευταία φάση αυτής της προγραμματικής περίοδου το θέμα της χρηματοδότησης από μέρους της Ιταλίας. Η κυρία Βαντερ Λάιεν έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό που μπορώ να σας πω είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις αρχίσουν να δέχονται, να λαμβάνουν οδηγίες από μέρους της Προέδρου Βαντελάιν, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα, θα επεξεργαστούμε τα θέματα αυτά. Πρόκειται για θέματα που αφορούν τις δαπάνες, προϋπολογισμό και βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι πολύ γρήγορα όλα αυτά θα τροφοδοτήσουν και τις διαπραγματεύσεις του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε μια ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση. Κυρία Γκίζε, αναφερθήκατε στις περιοχές που έχουν ανθρακοριχεία. Ναι. Αυτό βεβαίως αποτελεί τμήμα της εργασίας που θα αφορά αυτήν την μεταβατική χρηματοδότηση. Κύριε Πρόεδρε, η θέση της DG δεν μπορώ εδώ να παραπονεθώ για κάτι, γιατί η Γενική Διεύθυνσή μας μέχρι πέρσι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εργασίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό είναι κάτι που άλλαξε πέρσι. Αυτό εμπλούτησε τις σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε, ευελπιστούμε και προσδοκούμε πολύ ξεκάθαρα να παραμείνουμε σε αυτήν την θέση και να μπορούμε να συνεχίσουμε άσχετα με τον προγραμματισμό να επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις ε, σημαντικές διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν όσον αφορά την ανάπτυξη των περιφερειών. Εξαιτία της κρίσης μέχρι τώρα το σύμφωνο σταθερότητας, ανάπτυξης, τα προβλήματα εξοικονόμησης και λιτότητας ε, κυριαρχούσαν μέχρι τώρα, όμως είδαμε ότι οι επενδύσεις πλέον έχουν γίνει η κεντρική πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι αυτή η σημασία των επενδύσεων θα παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά για τις απαντήσεις σας, πολύ λεπτομερείς απαντήσεις προς τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι όλες οι απαντήσεις σας είναι εξαιρετικά χρήσιμες για μας, για την προετοιμασία του ή της υποψήφιου επιτρόπου. Διαθέτουμε σήμερα πληροφορίες και στοιχεία που θα μας επιτρέπουν να προετοιμάσουμε την ακρόαση αυτή. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι λάθη και σφάλματα θα πρέπει να αποφύγουμε βασιζόμενοι σε προηγούμενες προγραμματικές πολιτικές και στρατηγικές και δώσετε απαντήσεις σε πάρα πολλά από τα ερωτήματά μας, τα οποία σαφώς θα μας χρησιμεύσουν. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Περιμένουμε το Συμβούλιο για να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος με την Επιτροπή και ελπίζω πραγματικά ότι θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα πριν το τέλος του 2019. Αυτό όμως σημαίνει και προϋποθέτει ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη του το αποτέλεσμα προηγούμενων τριμερών διαλόγων. Γιατί υπάρχουν αποτελέσματα από τους τριμερείς διαλόγους του παρελθόντος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε στο προσδεκόμενο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας λέω στο επανειδήν. Και φτάσαμε και στο τέλος της συνεδρίασής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά όλους για τη συμμετοχή σας από το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, μια πλούσια συζήτηση, δυναμική συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 2 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί, καθώς και στις 3 Οκτωβρίου. Θα συνεδριάσουμε την Δετάρτη και την Πέμπτη, 2 και 3 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, οι οποίοι μας βοήθησαν να έχουμε υψηλής ποιότητας συζητήσεις.